Bene, allora cominciamo, anche perché poi oggi abbiamo la presenza. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο Λιθουανούς ε, υπουργούς και κατόπιν ε, θα εξετάσουμε ε, θα έχουμε τη συζήτηση με την Επίτροπο, κυρία Κρέσ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καλωσορίσουμε στην Επιτροπή Ήτρε, τον Επίτροπο κύριο Γκούστας, ο οποίος ε, είναι Επίτροπος, ε, μάλλον υπουργό Οικονομίας, ε, κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας. Και νομίζω ότι στην Επιτροπή Βιομηχανίας θα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να συναντηθούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή μας ε, θα επισκεφτεί το Βίλνιους και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ε, κύριε Υπουργέ, σας δίνω το λόγο και μετά οι συνάδελφοι θα έχουν δυνατότητα να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου προσφέρετε την ευκαιρία να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας ε, τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 500 εκατομμυρίων ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λιθουανική Προεδρία κατανοεί πλήρως ε, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζεται ε, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ε, Προεδρίας μας ε, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην ε, ανάπτυξη και στο άνοιγμα της Ευρώπης. Κατά τους επόμενους έξι μήνες θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις επικοδομητικές συναντήσεις με άλλους θεσμούς έτσι ώστε να επιτύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρώπης ως ε, ένας ε, αμερόληπτος ε, διαμεσολαβητής η Λιθουανία θα προσπαθήσει να προάγει τις συμβουλευτικές διαδικασίες που θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δράτομαι λοιπόν τις ευκαιρίες για να συγχαρώ την Ιρλανδική Προεδρία για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει κυρίως στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα. Η σημερινή ευκαιρία αποτελεί πολύ καλή, ε, η σημερινή συνάντηση αποτελεί πολύ καλή ευκαιρία για μένα να συναντηθώ μαζί σας γιατί με ενδιαφέρει να συνεργαστούμε καλά και θεωρώ ότι θα ωφεληθώ. Ε, ξεκινάμε λοιπόν με θέματα βιομηχανίας, καινοτομιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ε, η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία προσπάθησε να επιτύχει την ανάκαμψη. Αυτή η προσπάθειά μας ε, ήταν ε, σαφής. Για να μπορέσουν όμως οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να κατορθώσουν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης, είναι απαραίτητο για εμάς να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε σωστή βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και επιθυμώ να διασφαλίσω ότι η δική μας η Προεδρία θα εστιάσει την προσοχή της στην ε, εφαρμογή ανταγωνιστικών, ανταγωνιστικής βιομηχανικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, να επιτύχουμε πρόοδο και επίσης ε, χρειαζόμαστε να δούμε τι άλλες βελτιώσεις μπορούμε να σημειώσουμε για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και να ε, συμφωνήσουμε σχετικά με τις βράχοι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες που είναι η στήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. να τονώσουμε τη ζήτηση για τις υπηρεσίες ε, και τα εμπορεύματα και επίσης ε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση ανταγωνιστικότητας. Όσον αφορά την πρόσβαση ε, στις, στις δεξιότητες, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορέσουν να ε, επεκταθούν περαιτέρω. Ως πρώτο βήμα προτιθέμεθα να προάγουμε την καινοτομία μέσα από τις ε, δημόσιες ε, επενδύσεις. Εξάλλου θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τη βιομηχανική πολιτική στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας το Σεπτέμβριο. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας το Δεκέμβρη. Θα συνδυάσουμε την ανταγωνιστική πολιτική με την πολιτική βιομηχανίας και θα θελήσουμε επίσης να προάγουμε ε, τις ε, νέες καινοτόμες επιχειρήσεις ε, και την ανάπτυξη. Ο στόχος, ε, στον, ο μας είναι να έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ε, πολιτική καινοτομιών που θα εφαρμόσουμε. Τα συμπεράσματα θα συμπεριληφθούν στην έκθεση περί ανταγωνιστικότητας το 2013. Και αυτή θα είναι η συνεισφορά μας στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο του 2014. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ε, σημαντικό θέμα και αναφέρομαι σε αυτό που θα λάβει χώρα φέτος τον Οκτώβρη και θέλω να πω ότι η συμβολή στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, και αυτή θα είναι σημαντική και θα βασίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης των Καινοτομιών ε, και επίσης θα εμφανιστεί και στην ανακοίνωση σχετικά με το ρυθμό των καινοτομιών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κινητήρια δύναμη στην οικονομία μας και θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας θα έχουμε την πέμπτη επέτειο από την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις ε, θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή της αρχής ε, Think Small First και αυτό θα κυριαρχήσει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στο Βίλνιους. Το Σεπτέμβρη το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Βρυξέλλες θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των άτυπων συζητήσεων το αποτέλεσμα της ε, συζήτησης ε, για την πολιτική θα συμπεριληφθεί ε, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβρη. Ε, μας ενδιαφέρουν οι συζητήσεις για την εφαρμογή της ε, πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις. Επιθυμούμε να άρουμε όλα τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της πράξης αυτής. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσοχή ε, την σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είμαστε ευγνώμονες για τη δουλειά του κυρίου Ρούμπιχ σε αυτόν τον τομέα. Ε, στην συνέλευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, η οποία θα γίνει το Νοέμβριο στο Βίλνιο. Εκεί θα έχουμε εκπροσώπους ε, επιχειρήσεων οι εθνικές κυβερνήσεις και οι ακαδημαϊκοί θα συζητήσουν τη σημασία των εταιριών για την οικονομία και για την ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την κρίση. Επίσης ελπίζουμε οι συμμετέχοντες ε, να φύγουν από τη Λιτουανία με νέες απόψεις, επαφές και με ένα νέο όραμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή πρωτοβουλειών ε, καλύτερων ε, ρυθμίσεων που θα προάγουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες και ελπίζουμε αυτό να συμβάλλει στην ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Εξάλλου θα υπογραμμίσουμε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των υπαρχόντων εργαλείων όπως ε, τα τεστ, ε, οι δοκιμές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα προάγουμε τις βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη-μέλη και προτιθέμετα να αξιολογήσουμε το πώς ακριβώς το Συμβούλιο προτίθεται να συμπεριλάβει στην εργασία του και ε, ε, την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Όσον αφορά τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές αντιστοιχούν ή καταλαμβάνουν το 98% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η Ευρώπη θα ε, καταφύγει σε όλα τα μέτρα, έτσι ώστε να έχουμε την έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων ε, και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως από το 2014 και εφ' εξής. Τώρα, θα ήθελα να συνεχίσω με το θέμα της κόσμε και να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του προγράμματος αυτού. Ε, επιθυμώ να υπάρχει η ολοκλήρωση των ε, νομοθετικών ε, διαδικασιών. Όσον αφορά τώρα την πολιτική για το διάστημα. Κατανοούμε ότι η πολιτική αυτή θα έχει επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και της ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν στις νομικές πράξεις. Πρώτα απ' όλα επιθυμούμε πρόοδο ε, όσον αφορά την πρόταση Επιτροπής για το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Κατανοούμε τη σημασία αυτού του προγράμματος και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ε, δημιουργηθεί η νομοθετική βάση για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Έτσι λοιπόν ε, προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε πρόοδο για την απόφαση σχετικά ε, με το πρόγραμμα παρακολούθησης ε, και εντοπισμού, ε, διαστημικής παρακολούθησης και εντοπισμού. Στο Συμβούλιο θα διεκδικήσουμε την συνένεση για θέματα όπως πολιτική για τα δεδομένα, διακυβέρνηση και μηχανισμός χρηματοδότησης. Είμαστε ευγνώμονες στην εισηγήτρια, την κυρία Άντας Ντότα, για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος και προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία στο εγγύς μέλλον. Κατά τη διάρκεια της Λιτουανικής Προεδρίας θέλουμε να σας καλέσουμε, κυρία Πρόεδρε, να συμμετάσχετε στην διεθνή διάσκεψη με θέμα οικονομία διαστήματος στον πολυπολικό κόσμο που θα λάβει η χώρα στο Βίρνιο στις 18 έως 20 Σεπτεμβρίου. Αυτό θα είναι το τέταρτο συνέδριο, ένα από τα μεγαλύτερα στις χώρες της Βαλτικής, όπου ε, θα ε, συγκεντρωθούν διακεκριμένοι πυρογνώμονες από προγράμματα, από χώρες με διαστημικά προγράμματα. Εφέτος ε, η συνεδρίαση στο Βίλνιους θα οργανωθεί, θα λάβει χώρα από κοινού με την έκθεση για το διάστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βίλνιους. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ελπίζω ότι η μελλοντική μας συνεργασία θα είναι επικοδομητική, χρήσιμη και επιτυχής. Και θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και κυρία Πρόεδρε με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχουν τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε Υπουργέ για την εισηγησή σας αυτή. Ήταν διεξοδική για να δούμε τα ζητήματα που θα εξετάσουμε τους ερχόμενους μήνες. Να ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο Χίμπνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μας υπάρχουν κάποια θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το πώς θα προχωρήσουν στο Συμβούλιο. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε για τις δημοπρασίες ETS. Τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου ε, και το πώς όλα αυτά θα δημορφωθούν στην αγορά. 900 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται από την Προεδρία ότι θα αποκομίσουμε. Πιστεύετε ότι είναι καλό το ποσό αυτό για την βιομηχανία και σκοπεύετε να οργανώσετε συζητήσεις για τις αλλαγές στο σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών. Τι συνομιλίες θα έχετε με τα κάτι μέλη για το θέμα αυτό και με τους ευρωβουλευτές και για τις νησίδες ενέργειας όπως έχουν ονομαστεί. Ξέρουμε, ξέρετε ότι η Λιθουανία είναι μια περιοχή που δεν διαθέτει ενεργειακούς πόρους ε, συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε η μόνη περίπτωση ενεργειακή νησίδα στην Ευρώπη. Έχετε λοιπόν κάποια άποψη για το πώ αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα έπρεπε να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Χίμπνερ. Ο κύριος Μπαλσίτης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας, ε, συγχαρώ, και να σας ευχηθώ μάλλον κάθε, καλή, κάθε τύχη για αυτό το εξάμενο. Έχετε αναλάβει μάλιστα και το Υπουργείο αυτό και την Προεδρία ταυτόχρονα. Ασχολείστε με θέματα έρευνας, κοινοτομίας, διαστήματος, ε, και άλλους πολλούς τομείς που είναι σημαντικοί για τους ε, πολίτες μας. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις. Αναφέρατε στις δημόσιες προμήθειες. Όπως θα ξέρετε το Ευρωκοινοβούλιο συζήτησε το θέμα αυτό επανελειμμένος και το συζητάει εδώ και χρόνια και έχουμε καταλήξει σε πολλές συμφωνίες οι οποίες έχουν οδηγήσει στην έγκριση ψηφισμάτων με συγκεκριμένε διατάξεις. Προβλέπουν ότι ο τομέας των δημόσιων ε, αγορών θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πετύχει πολλά σε αυτό το τομέα η Λιθουανία. Έχει συγκεντρώσει αρκετή πείρα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς ε, στον τομέα των δημόσιων προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα επιτέγματα της Λιθουανίας και άλλων χωρών που θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστούμε Υπουργέ για την ε, παρουσία σας. Εδώ ήθελα να... Πάρω αφορμή από την αναφορά που κάνατε στο πρόγραμμα Κοπέρνικους. Είναι ένα πρόγραμμα άκρο σημαντικό γιατί είναι στην εμπροστοφυλακή στην αιχμή της τεχνολογίας και χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη και καλά μελετημένη διαχείριση της, ε, της εδαφικής διάστασης, αναλαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, αλλά και τις διοικητικές πρακτικές που έχουν σχέση με την γεωργία. Ε, έχει να κάνει με τη διαχείριση της γης και του εδάφους δηλαδή, με δυνατότητα ε, πολύ προηγμένων ε, μέσων, χρήσης προηγμένων μέσων. Πώς διασυνδέεται το πρόγραμμα αυτό με, το, με την άλλη υποδομή του προγράμματος Γκαλιλαίο. αυτό μπορεί να μας δώσει μια πολύ συγκεκριμένη γεωγραφική, ένα πολύ γεωγραφικό εντοπισμό, συγκεκριμένο γεωγραφικό εντοπισμό της σημερινή κατάστασης με το GPS. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη και μάλιστα μελητή, ότι τα ποσά που προβλέπονται για χρηματοδότηση ήδη έχουν ε, ε, πάρει την πορεία τους και θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα συγκεκριμένο ρυθμό για τις δαπάνες. Δεν θέλουμε να χαθεί άλλος χρόνος. Και επιπλέον γιατί θεωρώ ότι αυτό το εργαλείο είναι καθοριστική σημασίας για να διαχειριστούμε με τρόπο αποτελεσματικό και τις πολιτικές ε, καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και τις πολιτικές προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, νομίζω και θεωρώ ότι μπορούμε και οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια ταχεία υλοποίηση. Και γιατί έτσι θα εκμεταλλευτούμε το δυναμικό για την ε, εκπαίδευση των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την διαχείριση του εδάφους. Θα ήταν ε, πολύ σημαντική συμβολή τους και για τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν μέρου του Ευρωπαϊκού Κόμματο, κύριε Υπουργέ, σα ευχόμεθα. Καλώ ορίσατε στο Κοινοβούλιο. Δηλώνω με πρόθυμη να συνεργαστούμε μαζί σα. Η χώρα την οποία προέρχεστε έχει 20% βιομηχάνηση. Δηλαδή είστε κάτω από τον μέσο όρο που έχει τάξει. Συγγνώμη, πάνω το μέσο όρο που έχει τάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 16%. Εγώ εξέλεγε σε χώρα που αποβιομηχανοποιείται. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε να αναλύσουμε ποιο είναι το μυστικό της χώρας σας. Τώρα, κάτι άλλο. Όταν συζητήσαμε με τον πρώτο της Δημοκρατίας, συζητήθηκε το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία, διότι με την πολιτική γειτονία τη δεν περιλαμβάνουμε τη Ρωσία. Μόνο πείτε δύο λόγια, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι φυσικό συνομιλητή, φυσικό εταίρο τη Ένωση η Ρωσία. Θεωρείτε ότι πρέπει να συνάψουμε και βιομηχανικέ σχέσει με τη Ρωσία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Να δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό. Στον Υπουργό για τις πρώτες του απαντήσεις. Και έπειτα βλέπουμε αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις για να απαντήσετε. Visų pirma, noriu λέει ο Υπουργός Γκούστας Σα ευχαριστώ που θέσατε αυτές τις ερωτήσεις. Και ήθελα επίσης να σε ευχαριστήσω για την υποστήριξη την οποία μας προσφέρετε γιατί θα την χρειαστούμε κατά το εξάμεινο θα ασκήσουμε την Προεδρία βεβαίω και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τρόπο αποτελεσματικό. Σα ευχαριστώ όμω εκ των προτέρων. Τώρα, για το ETS και την αναβιομηχάνηση, ανα, την εκβιομηχάνηση τέλος πάντων εκ νέου της χώρας μας. Είναι κάτι βέβαια το οποίο άρκετα είναι με την οικονομική ανάπτυξη που γνωρίζει η χώρα μας. Πράσινη οικονομία προσπάθεια συγκράτησης του φαινομένου της αναθερμανίας του πλανήτη. Αυτά και τα δύο αποτελούν μεταβλητές που επηρεάζουν την βιομηχανία, διότι το κόστος της βιομηχανικής παραγωγής αυξάνεται. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αναγκάζεται η βιομηχανία να αγκαλιάσει καινοτόμε λύσεις. Άρα θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία. Ελπίζουμε ότι αυτή την ισορροπία θα την πετύχουμε θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο των διαπραγματεύσεων, την αναζήτηση συνένεσης στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε για τα όσα είπατε. Ναι, αποτελούμε ενεργειακή νήσο. Επίσης, Νομίζω ότι χθε ο σάνθος μου που σας μίλησε σας εξήγησε τις προτεραιότητες μας, αλλά μπορώ και να σα επαναλάβω ότι θέλουμε την ανάπτυξη και ε, ολοκλήρωση τη ενεργικής αγοράς. Έχουμε ως ορόσημο το έτος 2015. Επίσης, τη διασύνδεση της τους αγωγούς μεταφοράς της ενεργείας. Επίσης. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε ο κ. Μπαλτσίδης όσον αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες και διαγωνισμούς. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όσον αφορά τις ε, συμβάσεις και τους διαγωνισμούς, η χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε αυτή μας την ε, εμπειρία στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού ή ανταγωνιστικότητα του Ιουλίου. Να δούμε ακριβώς πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο έχουμε το 80% αυτών των συμβάσεων και διαγωνισμών που γίνονται ηλεκτρονικά. Μια επίδοση αξιόλογη. Επίσης σας τονίζω ότι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι το να μπορέσουμε να πετύχουμε και στο μέτωπο της καινοτομίας όσον αφορά τη συμβάση και του διαγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε οδηγηθεί στην ηλεκτρονική μέθοδο. Έχουμε δει ένα 10% του ΑΕΠ που πηγαίνει εκεί σε αυτές τις προμήθειες και μιλάμε για 420 δις. Πάρα πολύ, τεράστιο ποσό. Επομένως θα πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα με την ηλεκτρονική μέθοδο. Και για αυτό το λόγο και περιμένουμε πώς και πώς μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά ε, την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για αυτού τους λογαριασμούς. Θα γίνει ε, σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο και θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί πρόοδος και σε αυτό το μέτωπο κατά την Λιθουανική Προεδρία. Κύριε Πρόντι, ρωτήσατε για τον Κοπέρνικο, το πρόγραμμα Κοπέρνικος και έχετε δίκιο. Ανέφερα στην εισήγησή μου ότι η πολιτική του διαστήματος θα είναι μια μας προτεραιότητα. Και με το πρόγραμμα Κοπέρνικος θα συμβάλλουμε στην παρατηρήση της ε, υδρογείου. πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Κοπέρνικο και για θέσει απασχόληση και για την οικονομία γενικότερα, ειδικότερα για τις ΜΜΕ. Αυτό για μα είναι σαφέστατο. Επομένω και εμεί θα καταβάλουμε πάσα προσπάθεια ούτω ώστε εγκαίρω να εγκριθεί η σχετική νομοθετική πράξη, το σχετικό νομοθέτημα, ούτω ώστε να γίνει λειτουργικό και επιχειρησιακό το πρόγραμμα κοπέρνικο από το έτος 2014. Όμως θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά την υπαρκή πρικοδότηση για το Κοπέρνικος, όπως γνωρίζετε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει κλείσει, έχει συμφωνηθεί. Οπότε έχει συζητηθεί και η πρικοδότηση του προγράμματος Κοπέρνικος. Σίγουρα είναι θετικό το ότι το μεγαλύτερο ποσό της χρηματοδότησης πρόκειται να διατεθεί στην αρχή του προγράμματος, του πολυετούς. Άρα θα τρέξει εύρυθμα το Κοπέρνικος, αλλά βέβαια θα πρέπει να γίνει σωστή απορρόφηση και χρήση των διατεθειμένων πόρων. Για τον κύριο Οντίτορ. Έχετε δίκιο, κύριε Οντή. Η βιομηχανία γεννά 24% του ΑΕΠ μας. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε από 24% στο 25%. Έχουμε βέβαια και την πρόταση του ή Αντιπροέδρου της Επιτροπής για την αναβιομηχάνηση. Για να πάμε στο 20% σαν μισό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να κατέβουμε για να φτάσουμε αυτό τον δίκτυο. Αλλά να. Τι να σας πω για τη συνταγή επιτυχία μας. Δύσκολο να σας απαντήσω. Έχουμε χημικά, έχουμε ξυλία, είδη διατροφής, έπιπλα, σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε αναπτύξει μηχανία και διαθλητισμό και πασχίζουμε να κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα η βιομηχανία μας. Επίσης, έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε για την Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει περιληφθεί στην πολιτική την της Ανατολάς. Όμως, δεν έχουμε σχέσεις. Άλλες ε, ε, και εξαγωγές και εισαγωγές έχουμε με τη χώρα αυτή. Βεβαίω θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τη σχέση μας με τη Ρωσία. Και νομίζω θα είναι κάτι θετικό εάν συσφίξει τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Πολύ ωραία λοιπόν, ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, έχουμε μία ακόμα ερώτηση και κλείνει ο κατάλογος ε, από, τον, από τη συνάδελφο Μπαρέα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Δύσκολο, πρόεδρε, όπως προείπατε. Η επαναβιομηχάνηση, το μέλλον της βιομηχανίας, αυτό είναι το, είναι το μέλλον των ε, που θέλουμε στην Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και το ε, Συμβούλιο της Συνταγωνιστικότητας για ανταγωνισμό που περιμένουμε να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις αλλά χωρίς προϋπολογισμό πολιτική δεν ασκείται και έχουμε πρόβλημα έχουμε λιτότητα στα δημοσιονομικά Εντάξει, όπως είπατε έχουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο του 1997. Από παντού έχουμε απώλειες. Πρόβλημα στην πίστοση. Ε, τα επιτόκια είναι πρόβλημα. Άλλοι ε, δανείζονται με 0,5% και η Ισπανία με 8%. Τι θα κάνετε, τι μέτρα μπορεί να λάβετε τόσο ώστε να κλείσει το χάσμα μεταξύ μέρους χωρών. Πώς θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε, να γεφυρώσουμε. Το θέμα. Τελειώσαμε λοιπόν και κατόπιν τούτου κύριε Υπουργέ ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απαντήσετε σε αυτήν την τελευταία ερώτηση της ε, συναδέλφου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι η εκβιομηχάνηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Τώρα, ε, ως προς το τι προγραμματίζουμε κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας, όπως ίσως ε, θα έχετε παρατηρήσει στο πρόγραμμα της Προεδρίας αλλά και το δικό μου το σημαντικότερο όλων είναι να υπάρχει μεγαλύτερος, ε, περισσότεροι κανόνες στη βιομηχανική πολιτική και να υπάρχουν και διατάξεις ε, για τις ε, συστάσεις. Όπως σας είπα, τον Ιούλιο στο άτυπο συμβούλιο θα μιλήσουμε για αποτελεσματικότητα, για δημόσια επιχειρήσεις, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ηλεκτρονικές προμήθειες και επίσης ε, θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και αργότερα. Και ελπίζω ότι το Δεκέμβρη, αφού θα έχουν ακουστεί όλες οι προτάσεις και οι απόψεις, συμπεριλαμβανομένης και της ανακοίνωσης της Επιτροπής, τότε θα κατορθώσουμε να καταθέσουμε συμπεράσματα που θα μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια πολύ καλή συζήτηση για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Εμείς αναζητούμε πρόοδο σε αυτό τον τομέα. Τώρα, ε, σχετικά με το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι μικρότερο από ό,τι περιμέναμε στον τομέα της ε, ανταγωνιστικότητας και ε, υπάρχει σίγουρα ένα κομμάτι που αφορά τον εκβιομηχανισμό, όμως ο προπολογισμό δεν είναι ο καθοριστικός παράγων για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και όπως σας είπα, πρέπει να αναθεωρηθεί η νομική βάση, διότι βλέπουμε να υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα με την τρέχουσα νομοθεσία. Θέλω επίσης ε, να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να προάγουμε καινοτόμε πολιτικές όπως την αυξημένη ζήτηση για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την προαγωγή των ε, συγκεντρωτικών ε, σχημάτων, των δικτύων, ε, καλύτερη αξιολόγηση επιπτώσεων. Νομίζω λοιπόν ότι ο προπολογισμός είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι και ο καθοριστικός. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούν να προ... Πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσία σας, ε, για τη διαθεσιμότητά σας και άλλη φορά ε, θα σας φιλοξενήσουμε με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχόμαστε καλή δουλειά κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας. Επίσης ε, θα λάβουμε υπόψη μας τις ε, προτάσεις σας και χαίρομαι ε, για τη συνεργασία κατά τους επόμενους 6 μήνες. Possiamo cominciare il... Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ως ε, Επιτροπή Ήτρε θέλουμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντάνης Παλβάκη ε, που είναι υπουργό Παιδείας και Επιστημών της ε, Λιθωνικής Προεδρίας θα μείνει κοντά μας ε, για τα επόμενα 50 λεπτά ε, και θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας για τα δικά του τα θέματα και βέβαια μετά θα έχουμε και τη σχετική ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές προσκεκλημένη. Για μένα αποτελεί μεγάλη τιμή, προνόμιο. Είναι επίσης μεγάλη μου ευχαρίστηση και παράλληλα μία πρόκληση να σας μιλήσω σήμερα και να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Θεωρούμε ότι η Προεδρία μας θα δραματίσει σημαντικό ρόλο. Και με αυτή την ευκαιρία θα συνεχίσουμε το διάλογο και τη συνεργασία μαζί σας εκμεταλλευόμενοι την καλή σας διάθεση. Έχουν περάσει δύο εβδομάδε, ήταν τόσο σημαντική η διοργανική συμφωνία που αφορούσε την επιτυχιακή συμφωνία για το πρόγραμμα Horizon 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο και εργαλείο αυτό, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση και να μπορέσουμε να αλκίσουμε κορυφαίους ερευνητές, όπως επίσης και επιχειρήσεις καινοτόμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θετικό βήμα, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, τα μέλη της Επιτροπής, γιατί έχουν παίξει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για το πρόγραμμα 2020 ορίζον 2020 και επίσης θέλουμε να συνεχιστεί για την ολοκλήρωση της διαδρομής και συνεργασία μαζί σας. Επίσης θέλω να συγχαρώ την προηγούμενη Προεδρία, την Ισλανδική Προεδρία για το τιτάνιο έργο το οποίο επετέλεσε και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την επίκριση των στόχων που έχουν ε, συμφωνηθεί για τα πλαίσια της Τρόικα με και Ελλάδα. Κατά την Προεδρία μας επίσης θα, μπορούμε, δούμε πώς είναι δυνατόν να δούμε για το πώς μπορούμε να έχουμε τίμιο και αντικειμενικό ρόλο ως διαμεσολαβητές ε, ή στον διάλογο Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψη απόφασης έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς έχουμε δεσμευθεί ούτως ώστε να έχουμε αυτήν την επικοδομητική στενή συνεργασία μαζί σας. Όλα αυτά προς όφελος των Ευρωπαίων. Φέτος είναι το έτος του Ευρωπαίου πολίτου και θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπαθειές τους ούτως ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούν από εμάς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί σίγουρα τους αξίζουν καλύτερα, τους αξίζουν καλύτερες προοπτικές. Αυτό είναι βέβαιο. Κατά τις προετοιμασίες για την Προεδρία μας, είχα την ευκαιρία να συναντήσω την Πρόεδρο της ε, Επιτροπής σας, την κυρία Σαρτόρη. Την Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας Ερεύνης και Ενεργείας, αλλά και τον κύριο Έλερ, όπως και άλλα μέλη της Επιτροπής. Σε μια εβδομάδα επίσης πρόκειται να υποδεχθούμε την αντιπροσωπεία σας ή στο Βίλνιους. Όλα αυτά ελπίζω ότι θα βοηθήσουν ούτως ώστε να υπάρξει αλληλοκατανόηση και προσπάθεια για τους κοινούς στόχους. Η Λιθωνική Προεδρία θα έχει ως βασική προτεραιότητα την έρευνα και οπότε θα αρχίσουμε το 2014 την ε, πρόθεση του προγράμματος Ορίζον 2020. Καταρχήν υπήρχε συμφωνία όσον αφορά το νομοθετικό πακέτο για το πρόγραμμα αυτό. Οπότε θα πρέπει όμω ακόμη να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα. Επίσης, η Προεδρία πρόκειται να αναζητήσει τις σωστές λύσεις για το πρόγραμμα της Ευρατόμ και επίσης ε, να συμβάλλει ως Ευρώπη ή στο διεθνές ε, πρόγραμμα ITER ε, για την σύνδεξη. λάβαμε υπόψη φυσικά για το πρόγραμμα του 2020 την εκδέσή σας. Βέβαια. Έχουμε το άρθρο 85 της συνθήκης, βάση του οποίου θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την, ε, στην συνεργασία μας. Άλλο ζήτημα σημασίας για όλους μας είναι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας το 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση. Αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τον χώρο αριστείας και ανάπτυξης και έρευνας. Φέτος πρόκειται να έχουμε την πρώτη έκθεση πεπραγμένων έκθεση πρόοδου. Και τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, οι προτάσεις σας και οι παρατηρήσεις σας, αλλά και οι ερωτήσεις σας, πρόκειται να ζητηθούν κατά την διάσκεψη που θα οργανώσουμε στη Λιδονία. Προσωπικά θα ασχοληθώ, θα είμαι εκεί, οπότε και οι παρατηρήσεις σας πρόκειται να διαβαστούν εκεί που πρέπει. επίσης σας αναφέρω μόνο μόνο το ότι σε αυτή τη διάσκεψη θα συζητήσουμε την αναβάθμιση της ε, συνεργασίας μας, ε, της συνεργασίας μας προς Ανατολάς. Θα έχουμε ανθρώπινους πόρους, ε, οριζόντες για κοινωνικές επιστήμες αλλά και ανθρωπιστικές επιστήμες, FISA 13, Jurad Waste 13, το Φόρουμ της Καινοτομίας και άλλες επιμέρους διασκέψεις. Θα έχουμε δύο επίσημα και ένα ανεπίσημο συμβούλιο. Το επίσημη συνάντηση θα γίνει σε 15 μέρες στο Βίλνιος. Εκεί θα συζητήσουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα του τι δεξιότητες, τι παιδεία χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όσα απαιτούν οι καινοτόμε τεχνολογίε στην Ευρώπη. Γιατί ακόμα υπάρχει α, ασυμφωνία, αναντιστοιχία μεταξύ του τι πρέπει να κάνουμε και τι δάσκουν τα πανεπιστήμια. Επομένω, σε συναντήσει και στι Βρυξέλλε και στην Λιθουανία. Κυρία Σαρτόρη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Τελειώνει. Σε λίγο ε, που κοινοβηθεί αυτή η θητεία. Και βεβαίω ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού να ολοκληρώσουμε διαπραγματεύσει σε όσο γίνεται περισσότερα νομοθετήματα και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε όσο γίνεται πιο στενά με τους συνομοθέτες. Το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας και ενέργεια εκεί που το χαρτοφυλάκι μου ε, επιβάλλει τη συνεργασία. Και στην αρχή της ε, Προεδρίας σας είπα ότι θέλω να συνεργαστούμε το δεύτερο εξάμεινο και την επόμενη να τα στο Βίλνιος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τώρα τις ερωτήσεις σας, τις οποίες θα διαβιβάσω στις συναντήσεις, στα συμπόσια, στις διασκέψεις που θα κάνουμε στην Πληθωνία. Ευχαριστούμε, Υπουργέ να ξεκινήσουμε με του συναδέλφου και την κυρία Πιλάρ Τελκαστίγιο, εκ μέρου του ΕΛΚ. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Φορές τα ακουστικά σας και τώρα θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα ισπανικά. Καλώς ορίσατε από το Λαϊκό Κόμματο στην Επιτροπή μα. Όπω μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε αρμοδιότητα για θέματα έρευνα και καινοτομίας. Οπότε και μετά φυσικό είναι να ασχολούμεθα με το σχετικό πρόγραμμα Μάρκο και τα έγγραφα. Πώς, πώς, ακούτε την μετάφραση. If not, I can use English, but you don't... Αν έχετε πρόβλημα με τη μετάφραση, να σας τα πω στα αγγλικά. Άρα τα παραλαμβάνω αυτά που είπα. Και παραλαμβάνει η ομιλήτρια. Καλώς ορίσατε στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή. Εμείς έχουμε την ε, αρμοδιότητα για έρευνα και καινοτομία για το πρόγραμμα πλαίσιο. Επιμέρους, πιο συγκεκριμένα προγράμματα. Για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας. Όλα αυτά τα στοιχεία που καλεί το πρόγραμμα πλαίσιο του προγράμματος ορισμού 2020. Και το Κοινοβούλιο ασχολείται με αυτά τα θέματα, όχι μόνο όταν αυτά τα κατεβάζουν προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πριν, πριν από αυτήν. Όπως ας πούμε, τη θέμα της απλοποίησης, της διευκόλυνσης της συμμετοχής και αυτό, το θέμα αυτό εδώ με την ε, συνάδελφο Παρβάλλο το συζητήσαμε εδώ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ιρλανδική Προεδρία. Αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή και την Επιτροπή για αυτά τα οποία έκανε, που έκανε προσπάθεια εξαιρετική. δύσκολα θέματα, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Δηλαδή, πολλές φορές κάτι θα πρέπει να προσθέσει κανείς, να αλλάξει μια λεξούλα εδώ, μια λεξούλα εκεί. Οπότε και δεν μπορώ παρά να σας ζητήσω, μια που εκπροσωπείτε την τηλεφωνική ε, Προεδρία, να καταβάλλετε ό,τι προσπάθεια μπορείτε ούτως ώστε όλες αυτές οι λεπτές, οι δύσκολες λεπτομέρειες να διευκρινίζονται, να λύνονται τα προβλήματα. Ότι κρεμοί να διεκπαιρεώνται όσο γίνεται πιο γρήγορα Και βέβαια είναι το θέμα της ε, έρευνας το οποίο θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε γι' αυτό. Ένα άλλο μέτωπο είναι μια προσπάθεια στην οποία, την οποία πρέπει να καταβάλλετε. Κάτι να κάνετε για αυτό το θέμα, γιατί οι Ευρωπαίοι ερευνητέ περιμένουν πώς και πώς να κάνουμε κάτι. Γιατί άλλωστε υπάρχει πρόβλημα με τα κονδύλια τα οποία αφορούν την ε, έρευνα. στι περισσότερες χώρες είναι προφανές γιατί είναι λόγω της κρίσης. Οπότε, σαν το μάνα εξ το περιμένουμε. Να υπάρξουν οι αναγκαίοι πόροι για τα ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι τα επανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα να μπορέσουν να καλυφθούν με αυτούς τους πόρους που τόσο τους χρειάζονται. Άρα, το νωρίτερο δυνατόν. Κλείστε ό,τι συμφωνία χρειάζεται να κλείσετε και διαθέστε όσο γίνεται μεγαλύτερη επικοδότηση. Και να ξέρετε ότι όποτε έρχεστε εδώ πάντα θα είστε ευπρόσδεκτος. Πιλάρης ευχαριστώ. Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί είναι η τρίτη φορά που ζητώ το λόγο σήμερα και τον παίρνω. Διότι είναι ο τρίτος υπουργό που υποδεχόμαστε στην Επιτροπή Ήτρε και θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να σας καλωσορίσω. Οι προεδρεύοντε υπουργοί, ιδίω εσεί, ε, κύριε Υπουργέ, έχετε αναλάβει ένα θέμα με πολλές Διαφορετικέ συνιστώσεις. Είστε επιστήμονα και εσεί ο ίδιο και γνωρίζετε πολύ καλά τι προκλήσει αυτέ. Και ήθελα να σα κάνω μία ερώτηση που αφορά συνολικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα των κλάστερ, των συνεργοτικών ομάδων που έχουν αναφερθεί ως ε, ένα τομέα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί χρειάζονται τεράστιε επενδύσει και έχουν γίνει στο παρελθόν σε πολλά κράτη-μέλη. Και μας ενδιαφέρουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί, τα κλάστερς και για τα κτίρια και για πολλούς τομείς ε, προτεραιότητας. Ξέρουμε ότι η διαδικασία του clustering ε, ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη και σε πολλούς τομείς σήμερα τα αποτελέσματα ακόμη δεν είναι ικανοποιητικά. Θα θέλαμε όμως να λάβουμε υπόψη και τα αισιόδοξα δείγματα. Πώς σκοπεύετε λοιπόν κύριε Υπουργέ να προχωρήσετε με πρωτοβουλίε σε αυτόν τον τομέα ώστε να δώσετε μια όθηση στον τομέα του clustering, να υπάρξει μια νέα πνοή ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τα επιστημονικά επιτεύγματα και να επιλύσουμε και προβλήματα που μπορεί να, έχουν, να κάνουν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλτσίτης και κυρία Καρβάλιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό στην Επιτροπή Ήτρε και να το ευχηθώ καλή τύχη για το επόμενο εξάμεινο, το εξάμεινο της Προεδρίας. Είμαι εισηγήτρια για το πρόγραμμα του Horizon 2020 και θα ήθελα να ενώσω τη φωνή μου με αυτήν της κυρίας Ντερκαστίγιο Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ όλα τα θεσμικά όργανα για την καλή συνεργασία που είχαμε και βεβαίως ε, το όργανο που εσείς εκπροσωπείτε, αυτό που, όπου συμμετέχουν δηλαδή τα κράτη-μέλη όπου μπορούν να βαρύνουν βεβαίως ε, στην διαμόρφωση του όλου προγράμματος. Η λύση νομίζω που βρέθηκε είναι αρκετά ισορρόπια, όπω η Συμφωνία για τις μικρομεσαίε επιχειρήσει, ο γενικό προπολογισμό, οι σχέση συνέργεια με τα διευθυντικά ταμεία και όπως είδα πρόσφατα σε δημοσιεύματα σε εφημερίδες, σχεδόν όλα τα πετύχαμε όσο θέλαμε για το πρόγραμμα αυτό, εκτός από τα κονδύλια, τον προπολογισμό. Θέλαμε μεγαλύτερα ποσά, Δυστυχώ δεν το πετύχαμε. Δεν μπορεί η έρευνα και υπεύθυνη έρευνα μόνο να καλύπτονται. Εάν το είχαμε καταφέρει και αυτό, το Horizon 2020 θα τα πήγαινε ακόμα καλύτερα, θα έχει ακόμα καλύτερε πιθανότητε από ό,τι έχει τώρα. Διότι τώρα ο προπολογισμό, όπω ξέρετε, δεν εκπροσωπεί πραγματικά αύξηση. Αύξηση, αν θεωρήσουμε βεβαίω όλα όσα συμπεριλαμβάνει το Horizon 2020. Όμως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ώστε όπως είπατε και εσείς Υπουργέ, να υλοποιήσουμε σωστά αυτά που απομένει να γίνουν ακόμη. Ιδίω προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα ξεκινήσουν γέρο στι αρχέ του 2014. Πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν, να περατωθούν τα κείμενα, ε, πολλή δουλειά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης, του Συμβουλίου, όμως ακόμη Κάποιες δράσεις όπως οι δράσεις υπό το άρθρο 1 και 5 με τη διαδικασία της συναπόφασης, τα EDCTP, η καταπολέμηση δηλαδή της ελονοσίας, της φυματίωσης και του AIDS, η δεύτερη φάση του προγράμματος δηλαδή. Όλα αυτά απαιτούν την έγκριση, δηλαδή την λήψη απόφασης και από το Κοινοβούλιο. Μόνον τότε θα καθοριστεί το ερχόμενο εξάμεινο, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα και να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα, ώστε όλα να είναι πλέον έτοιμα στο τέλος της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας επισκεφθείτε στην Επιτροπή μας θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Δύο σημεία. Πρώτον, για τους νέους. Είστε ε, υπουργός νεολε... της ε, παιδείας και συζητήσαμε για τα δημοσιονομικά κονδύλια αλλά και την κρίσιμη κατάσταση της ανεργίας των νέων. Συζητήσαμε τι πολιτικές θα χρειαστούν εδώ. Έχουμε ανάγκη από πολιτικούς μηχανικούς, από νέους επαγγελματικούς κλάδους, ιδίως για το cloud computing, το, τις νέες δηλαδή τεχνολογικές χρήσεις που έχουν να κάνουν με τις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας και ηλεκτρονικής. Θα πρέπει στα πλαίσια του προγράμματος 2000, για το 2020 να αναζητήσουμε νέες ιδέες, νέες ατραπούς. Υπάρχει εδώ κάποια τέτοια πρόθεση, γιατί θέλω να σας στηρίξω σε κάθε σχετική προσπάθεια. Πρέπει να γίνει μεγάλη, προσπά... μεγάλη πολλή δουλειά για τους νέους. Και έπειτα ένα δεύτερο σημείο που και εγώ συνεργάζομαι με τα πανεπιστήμια στην δική μου εκλογική περιφέρεια. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ε, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φτιαγμένες από φοιτητέ. Πώς τα ανώτερα στελέχη θα μπορούσαν να διευκολύνουν τους νέους ώστε να γίνουν οι νέοι ίδιοι επιχειρηματίες. Και ένα τρίτο σημείο Έχω μια ανησυχία, Υπουργέ, γιατί αυτό θα επισυμβεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Το τι γίνεται με τη στήριξη της κινητικότητας των νέων. Εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε θερμά υπέρμαχοι της κινητικότητα των νέων. Όμως δεν θέλουμε οι χώρες που ε, χρηματοδοτούν την εκπαίδευση, που επιτρέπουν ε, στους νέους να πάρουν διπλώματα, να είναι οι μόνοι ε, που λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις και ουσιαστικά αποστραγγίζουν από τους εγκεφάλους των νέων ε, τις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν την κινητικότητα των νέων, απλώς ανησυχώ λιγάκι. Ανησυχώ γιατί κάποιες χώρες για λόγους δημογραφικούς να προσελκύουν μαζικά νέους οι οποίοι μετά θα λείψουν από άλλες χώρες και για τις υποδομές. Συζητήσαμε για τα διευθυντικά ταμεία και διαπιστώνω ότι όλοι θέλουν να χρηματοδοτηθούν τα πάντα από τα διευθυντικά ταμεία. Εμεί δώσαμε αγώνα για να διατηρήσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε την έρευνα ε, από τα διευθυντικά ταμεία, τα χρειαζόμαστε για την ε, απασχόληση και για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Πώ βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα ω προ τον προπολογισμό, Έρχεστε από μια χώρα τη διεύρυνση, τουλάχιστον στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σα την άποψη για το πώ τα ταμεία αυτά, τα κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία μπορούν να, καθορίσουν, να διδαματίσουν καθοριστικό ρόλο στη σημερινή κατάσταση, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ισορροπία στους τομείς ενδιαφέροντο μα και κυρίω ε, στον τομέα του οποίου είστε υπεύθυνο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Εύαν. Κυρία Έλερ, συγγνώμη. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Δείξατε την ε, ιδιαίτερη σημασία που δίνετε στα θέματα αυτά και ότι ξεπερνάει τα όρια των στενών βιωτήτων της Προεδρίας σας. Θέλετε το Horizon 2020 να λειτουργήσει ως ε, ένα εμβληματικό στοιχείο του ευρωπαϊκού ε, του εξαμήνου σας και το ίδιο αισθάνεται και το Ευρωκοινοβούλιο. Μια ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι το Κοινοβούλιο προσέφερε συγκεκριμένα στη διαδικασία προσχώρηση της χώρας σας και προκειμένου να ωφεληθεί και η χώρα σας. Νομίζω ότι με την ε, βαθμίδα για την αριστεία έχουμε προσφέρει πολλά. Προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και βλέπουμε πλέον τα χειροπιαστά αποτελέσματα της προσπάθειας. Ευχαριστούμε και για τη δική σας τη στήριξη, διότι στην αρχή χρειάστηκε να πείσετε ολόκληρο το Συμβούλιο για το θέμα αυτό, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε μια κοινή ε, προσπάθεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Ακούσαμε διάφορε αναφορέ στα διευθυντικά ταμεία τον τον ε, κανονισμό για τα γεκλικά ταμεία κονδύλια και για, τον, για το Horizon 2020. Η βασική πρόκληση ποια είναι. Ότι ήταν χλιαρή η αντίδραση των κρατών μελών και στο να αποδώσουν κονδύλια για την ε, καινοτομία από τα διευθυντικά ταμεία και για την καινοτομία και για την έρευνα και για την εκπαίδευση και για όσα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν είναι σε τι βαθμό σκέφτεστε ή ετοιμάζεστε τι, ε, πώς το έδαφος για να ε, λάβουν όλα αυτά χώρα, να πάρουν σάρκα και οστά. Διότι τα κονδύλια των διευθυντικών ταμείων βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Μπορεί να μην αρέσει αυτό στα κρατημέλη, αλλά εδώ είναι. Εάν υπάρξουν λοιπόν περισσότερα κονδύλια, θα πρέπει να καθορίσουν τα κράτη-μέλη πώς θα τα χρησιμοποιήσουν θα τα χρησιμοποιήσουν αν θέλουν και την καινοτομία, αλλά μπορεί και όχι. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι χρειάζεται ώστε όλα αυτά να υλοποιηθούν, να γίνει απαραίτητη ε, σύνδεση μεταξύ των διευθυντικών ταμείων και του Horizon 2020. Και κατά δεύτερον, να σα ρωτήσουμε για τον προπολογισμό. Θα γνωρίζετε ότι σε πραγματικού όρου έχουμε περικοπή του 10%. Πάμε πάλι στα 70 εκατομμύρια. Ε, θα έπρεπε να είναι 77 για τι ανάγκε του 2013. Χοντρικά είναι 10% η μείωση αλλά ζούμε σε καιρούς οικονομικών προβλημάτων, δημοσιονομικής πίεσης, οπότε σε πραγματικούς όρους η επένδυση για το 2014 και 2015 θα πρέπει να παραμείνει παρούσα. Δεν θα μειωθεί όπως έγινε το 2013. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η προσπάθεια τουλάχιστον εντός Τη λεγόμενης ευελιξία να γίνει κάποια προσπάθεια ώστε το 2014 και 2015 να δαπανίσουμε τα πετούμενα κονδύλια σε καιρού και σε συγκυρίες μάλιστα κρίση. Υπάρχει μια προβλεπόμενη χρηματοδότηση μελλοντική και έπειτα για την ταχύτερη προσέγγιση, την ε, κατάντη προσέγγιση έχει να κάνει και με την υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία, εμπειρογνώμονες για να λειτουργήσουν όλα αυτά θα θέλατε λίγο να αναπτύξετε το πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της ταχείας διαδικασίας και να μας πείτε τι σημασία της δίνετε. Ωραία. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο. Εάν ικανοποιηθήκατε λοιπόν να δώσω το λόγο στον, το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με την εξής απάντηση. Κοιτάξτε, η ερώτησή σας μοιάζει με αυτή του κυρίου Έλα σχετικά με το fast track. Είναι του ιδίου στυλ και, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Ε, στο να εφαρμόσουμε ταχύτατα όλα αυτά που χρειάζονται. Από πλευράς ε, Συμβουλίου όμως ε, έχουμε καταθέσει επιτάπητος όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι περισσότερο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βεβαίως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο μπορούμε να δείξουμε ότι τώρα πια μπορούμε να προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι κατά το παρελθόν. Δηλαδή οι διαπραγματεύσεις να γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Γιατί ένα από τα αρνητικά στοιχεία ε, που συζητούνται γενικώ είναι ότι στις Βρυξέλλες υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό που ετέθη και υπήρξαν και άλλες δύο ερωτήσεις ε, σχετικά με την έλλειψη κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα θέλαμε για την έρευνα ε, και την καινοτομία να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια. Για έξι περίπου μήνες <coughs> επισκέφτηκα όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια, όλα τα πανεπιστημιακά φόρουμ για ανατεχνολογία και για πάρα πολλά άλλα θέματα και βασικά όλοι έλεγαν το ίδιο, ότι χρειάζονται κρίματα. Βεβαίω από την άλλη πλευρά Μόνο ε, σε αυτό το κονδύλι ε, του προπολογισμού δεν έχουν γίνει σημαντικές ε, περικοπές. Άλλα κονδύλια περικόπηκαν πολύ περισσότερο λόγω της κρίσης. Άρα δηλαδή αυτό είναι επίτευγμα και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι οι ερευνητές και όσοι ασχολούνται με την καινοτομία θα μας ευχαριστήσουν ε, για όλα αυτά. Και το έκανα και εγώ. Ο κύριος Μπαλτσίτης μου ζήτησε να σχολιάσω το θέμα των συνεργατικών σχηματισμών, των υποδομών και το ποια θα είναι τα επόμενά μας βήματα. Ελπίζω λοιπόν ότι η συνεργασία μας ε, οδήγησε στο να κλείσουν τα θέματα 187, 157 επίσης, 285 πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα ε, στους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να υπάρξουν ε, από κοινού προγράμματα στην καινοτόμο ιατρική, στην νανοτεχνολογία και σε άλλους τομείς, νομίζω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση της έρευνας και της τεχνολογίας και αυτή πρέπει να είναι ορατή. Γιατί όταν μιλάμε για έρευνα και καινοτομία, για το χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους, ξεχνάμε ότι μιλάμε για έρευνα που είναι ε, πολύ καλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρονται πολλές ιδέες και απόψεις σε τεχνολογική καινοτομία. Όμως εκεί που δεν είμαστε καλοί είναι στο να μεταφέρουμε την ε, παραγωγή στη βιομηχανία. Αυτό λοιπόν το κενό ε, πρέπει να καλυφθεί. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το αναγνωρίσουμε και από κοινού να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Κυρία Καρσία Κορβάλιο, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ε, σας λέω και πάλι ε, τέθη ένα πολύ σημαντικό θέμα σχετικά με τον ε, προϋπολογισμό και τα άρθρα 185 και 187. Η Λιθουανία θα εργαστεί σκληρά για να σημειώσει πρόοδο σε αυτά τα θέματα και μάλιστα αν μου επιτρέπετε, θα επανέλθω και αργότερα ε, για να κάνουμε τις απαραίτητες συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή. Κυρία Τράουτμαν, μας ε, έκανε ερωτήσεις ε, σχετικά με τους νέους, την κινητικότητα, την αφέμαξη εγκεφάλων και τον προϋπολογισμό. Και νομίζω ότι ε, για τον προπολογισμό έχω ήδη απαντήσει. Όσον αφορά τώρα την ανεργία των ε, νέων, αυτό νομίζω είναι πρώτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι συζητάνε για την ανεργία των νέων κατά την ε, τελετή έναρξης, ε, ανάληψης καθηκόντων της Λιθουανικής Προεδρίας. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν. Λέγοντας ότι οι νέοι δεν έχουν δουλειά, θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα σε αυτά που έχουν οι άνθρωποι και σε αυτά που είναι απαραίτητα, που χρειάζονται ε, στην ε, βιομηχανία. Έχουμε λοιπόν στην αγορά πολλού πολλούς άνεργους με κάποιες ειδικότητες και από την άλλη όμως ε, χρειαζόμαστε πολλούς ε, μηχανικούς ε, σε τομείς, σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που έδειξε η κυρία Τράουτμαν, που είναι πολύ σημαντικό. Και το τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε για το θέμα στο Vilnius θα συζητήσουμε για την απασχόληση και για το πώς θα μπορέσουμε να ταιριάξουμε τις δεξιότητες και τα προσόντα των πτυχιούχων ε, έτσι λοιπόν νομίζω ότι ε, θα αποκτήσουμε ε, κάποια θέματα, κάποια, κάποια θέματα Ο κύριος Έλλαρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Κοινοβουλίου ε, για το Horizon 2020. Τώρα, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, ε, θέλω να σας πω ότι επισκέφτηκα κάποιες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, προφανώς υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα ε, στην ε, διαρθρωτική εξειδίκευση και το ορίζον 2020. Επίσης, αναμφίβολα, θα μεριμνήσουμε στο να χρησιμοποιήσουμε διαρθρωτικά κονδύλια τα οποία θα επενδυθούν έτσι ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό όφελος και αποτέλεσμα για την κοινωνία, την καινοτομία και την ε, τεχνολογία. Η ερώτησή σας ε, λοιπόν είναι πολύ επίκαιρη και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το θέμα αυτό να ληφθεί περισσότερο υπόψη κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε Υπουργέ και για την προσελευσή σας και για την εισήγηση και για τις πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας λοιπόν σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και σας δίνουμε ραντεβού σε επόμενη ευκαιρία μέσα στο ερχόμενο εξάμενο για τις απαραίτητες ενημερώσεις. Σας ευχαριστούμε και στο επανεδίνη. Ξεκινούμε αμέσως, διότι έπρεπε να προσθέσουμε και ένα σημείο στη ημερήσια διάταξη. Το πρωί καθυστερήσαμε λιγάκι, οπότε δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στην συνάδελφο Χίμπνερ για να μας ενημερώσει για το COP19. το σημείο που μα έμεινε από το πρωί, των μέρων εθνών για την αλλαγή του κλίματο 2013. Μισό λεπτάκι να φύγουν οι συνάδελφοι από την αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη στα σχόλιά μου. Θα, θα σας μιλήσω για το θέμα που έχουμε ήδη καλύψει με τους κοιόδης συζητητές συναδέλφους μου. Ε, προ 15 συναντηθήκαμε και αποφασίσαμε να βασιστούμε στο έγγραφο που συντάχθηκε στην Επιτροπή πέρσι. Ήταν ένα ιδιαίτερα εύστοχο κείμενο και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη όλα τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν το έργο της Επιτροπής μας. Συγκεκριμένες προτάσεις τώρα τις έχω ε, ελέγξει και μελετήσει και κατέληξα ότι τρεις θα είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επικεντρώσω τα σχολεία μας για να δώσουμε τη σωστή έμφαση. Πρώτα απ' όλα ανταγωνιστικότητα και βιομηχανία, έπειτα έρευνα και κοινοτομία και έπειτα ενεργειακή πολιτική. Όλα αυτά όπως προέκυψαν και από την ε, Σύνοδο. Να πω λίγα λόγια για τα διαφορετικά, για τα επιμέρους κεφάλαια αυτά σε όλα προσπάθησα να δώσω γεγονότα, πιστήρια και επιστημονικά στοιχεία όσα έχουν προκύψει από την έρευνα ή από όσα ήδη έχουμε λάβει ως μέρος της ενημέρωσής μας. Και επιτά για το καθένα από τα κεφάλαια έχουμε αναφέρει τι θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει στην Σύνοδο. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα όπως προείπα, και θα πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι βάσει του εγγράφου και των δεδομένων που διαθέτουμε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, το 2012 αυξήθηκαν παρά την παράλληλη μείωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε κάνει λοιπόν ήδη διάγνωση, έχουμε προβλέψει ποιες είναι οι γεωγραφικές περιοχές του κόσμου που διωγγώνουν την, τον συνολικό όγκο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το επόμενο σημείο αφορά το εξή. Η κατανάλωση ενέργειας προφανώς θα αυξηθεί. Και αυτό λόγω της... και θα αφορά όλους τους ενεργειακούς πόρους μεγαλύτερη κατανάλωση όλων των ενεργειακών πόρων. Δεν θα φτάσει η μεγαλύτερη κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Καυσίμων που έρχονται από ανανεώσιμε πηγέ δηλαδή. Θα χρησιμοποιούνται τα καύσιμα στην Ευρώπη και στην αγορά τη Ευρώπη με πολλού διαφορετικού τρόπου. Εμεί θέλουμε σίγουρα να έχουμε μια ισόρροπη οικονομία για αυτό το σκοπό. Και θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονό ότι τα ανταγωνιστικά μα πλεονεκτήματα θέλουμε να τα διατηρήσουμε προκειμένου να υπάρχει ισόρροπη επαγγελματική και τεχνολογική γνώση. Σε τέτοιε συνόδου λοιπόν κορυφή για το κλίμα πρέπει να δούμε και να αναζητήσουμε τρόπου για να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το γεγονό ότι όλες αυτές οι προετοιμασίε για την σύνοδο καθορίζουν με τρόπο αρκετά αποφασιστικό και τις τιμές της ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τον αντίκτυπο των τιμών της ενέργειας, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη διάδοση κάθε είδους φιλική προ το περιβάλλον τεχνολογική λύση. Όπω λόγου χάρη των, των αποτελεσματικών, τη αποτελεσματική χρήση των ορυκτών καυσίμων ή την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εγκρίναμε το έγγραφο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το έγγραφο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ευρύτερο επίπεδο από ό,τι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ανά τον κόσμο. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από την πρότασή μας είναι το εξής και η βιομηχανία και οι καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμοι. Έτοιμοι να θέσουν φιλοδοξότερους στόχους για την κλιματική πολιτική. Όμως πιστεύουμε ότι το να γίνουν αποδεκτοί τέτοιου είδου στόχοι θα έχει πιθανότητες επιτυχίας μόνον εφόσον και οι υπόλοιπε ε, οικονομίες ε, ανά τον κόσμο κάνουν παρόμοιες προσπάθειες. Δεν μπορούμε να είμαστε ένας ε, μοναχικός, ένα καραβάκι που κλαίει μόνο του σε ένα τεράστιο ωκεανό. Ιδάλλω του στόχου αυτού μπορούμε να του ε, επιδιώκουμε μόνοι μα. Είμαστε μέρο μια ε, παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια προοπτική. Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει δείχνουν ότι οι εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνον είναι το 11% των παγκόσμιων εκπομπών, του όγκου των παγκόσμιων εκπομπών και θα μειωθούν, θα συρρυκνωθούν τις ερχόμενες δεκαετίες. Θα πρέπει λοιπόν να προειδοποιήσουμε και τους υπόλοιπους ε, ε, ανθρώπους στον κόσμο ότι είναι υπερφιλόδοξη η στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ίσως έτσι... Ε, μας ξεφύγουν οι εκπομπές, δηλαδή αν εισάγουμε προϊόντα από χώρες με μεγαλύτερο όγκο εκπομπών από ότι εμείς, μπορεί να αυξήσουμε και το δικό μας αποτέλεσμα. Ε, πρέπει να καλωσορίσουμε τις ενδείξεις που έχουμε λάβει και τα μηνύματα από τις ΗΠΑ που δείχνουν ότι υπάρχει θετικότερη στάση προς την ε, εξέβρεση μιας παγκόσμιας συμφωνίας. Βεβαίως, ε, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει και σε αυτή τη σύνοδο να επιδιώξουμε να συγκεντρώσουμε αυτό το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη, όχι μόνο από μικρές χώρες, αλλά από εκείνους που εκπέμπουν περισσότερο. Εκείνους που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει σε εκείνους να δώσουμε βάρος, ώστε να επιδιώξουμε από κοινού την επίτευξη κοινών στόχων. Όπως προείπα και τόνισα, καθένα από τα κεφάλαια θα είναι ε, ταυτόχρονα και μία έκκληση. Μία έκκληση που θα απευθύνεται σε όλους για στενότερη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που θα πρέπει να λειτουργήσει ε, με ιδιαίτερα ενεργό τρόπο να δραστηριοποιηθεί για να συμβάλλει στη σύνταξη τέτοιων κειμένων. Έχουμε και τους εθνικούς φορείς ενέργειας βεβαίως, τον Διεθνή Οργανισμό για τις Ανανώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εταιρική σχέση για την ε, συνεργασία και την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία με τρόπο ενεργό, ώστε να μην παραλείψουν το παραμικρό στοιχείο και να υπάρξει μια ισορροπημένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις νέες τεχνολογίες πάνω απ' όλα γνωρίζουμε ότι οι τεχνολογίες μπορεί να αποτελέσουν ε, ένα ορόσημο τη δυνατότητα να γίνει ένα δραστικό βήμα προς τις νέες τεχνολογίες και να ενθαρρύνουμε, να τονώσουμε τον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Δεν υπάρχει μόνο μία ή δύο λύσεις που θα μπορούσαν να ε, προωθηθούν, να προκριθούν και οι υπόλοιπε να διαγραφούν. Όχι όλες τις προσπάθειες υπέρ της καινοτομίας και της έρευνας που να τις στηρίξουμε και πρέπει να πείσουμε τους εταίρους μας από τον υπόλοιπο κόσμο να κάνουν το ίδιο. Ε, στην σύνοψη εδώ βλέπουμε έκκληση για παγκόσμια συνεργασία προκειμένου να, τονωθεί, να τονωθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Σήμερα Συζήτησα με ανθρώπους από το Silicon Valley για το τι πιστεύουν για τις εξελίξεις εκεί και για το μέλλον και πιστεύουν ότι θα υπάρξουν συστήματα που θα διασφαλίζουν την ενέργεια και θα αποτελέσουν πλέον τον κανόνα από, με λύσεις από το υπέδαφος, υπόγειες λύσεις. Μ, καταλαβαίνω δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να κλείσω. Για την ενεργειακή πολιτική. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιλήσουμε επιδοτήσεις ε, και να τις κατευθύνουμε σε αυτούς που δεν έχουν ακόμη προσαρμόσει τα τεχνολογικά τους μέσα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ο απλούστερος τρόπος για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μπορούν να συμβάλλουν στην αντιστροφή της τάσης για την ε, αύξηση και της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους και των τιμών. Μπορεί να, να διδραματίσει πολύ δραστικό ρόλο παγκοσμίω για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Πρόεδρος ευχαριστούμε. Αλλά καθώς πρέπει να κλείσουμε πριν από την άφηξη της Επιτρόπου και έχουμε ακόμη τρία θέματα, κάποια στιγμή θα αναγκαστώ να σας ζητήσω να σεβαστείτε αυστηρά τα χρονικά όρια. Τρία λεπτά λοιπόν στον συνάδελφο Σιμάνσκι, ε, επειδή είναι σκιώδης εισηγητής, και δύο λεπτά στους υπόλοιπους σκιώδης εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ, λέει Σιμάνσκι. Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ ότι πρόκειται απλώς για σχέδιο κειμένου και σχέδιο το οποίο βέβαια ε, θα το καταλάβουμε να ανοίξουμε μια ματιά στο ιστορικό των διαπραγματεύσεων αυτό το κοπ η Ρωσία, η Κίνα, η Βασιλεία είναι από τις όμορες οικονομίες και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Περιμένω τον τι θα κάνει η Ευρώπη. Τι θα γίνει με αυτούς τους στόχους που έχουμε τάξει και ανεξαρτήτως του ποιος ε, πρόκειται να μπει σε αυτήν την ε, ε, τεράστια προσπάθεια. Πάρα προσδοκία, παραπάσα προσδοκία, δεν κάνουν τίποτα οι βασικοί ανταγωνιστές μας. Μένω στα λόγια. Δεν είναι τίποτα. Και επομένω αυτή η 19 διάσκεψη μας ε, χτυπάει ένα καμπανάκι. Και έχουμε δε τα συμπέρασμα του 2007. Και άρα θα πρέπει να εξαρτάται οτιδήποτε άλλο κάνει στην από το εάν συμφωνείτε η συνεργασία, η σύμπραξη με κάποιον άλλο. Γιατί θα πρέπει να εξορροπήσουμε αυτούς τους φιλόδοξους ε, στόχους με τα σχέδιά μας, τα βιομηχανικά. Είδατε τι είπε πριν από δύο εβδομάδες η κυρία Μέρκελ μετά από κάποια συνάντηση του Συμβουλίου τότε που αποφάσισαν να μην ανέβουν τα όρια ε, εκπομπής διοξιδίου από τα καινούργια οχήματα. Στα αγγλικά, τι ε, μου εδώ πέρα κάθομαστε εδώ και μην συζητούμε για την απασχόληση. Ε, τα λέω στην αγγλικά για να γίνει λάθος. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επιβάλλεται η σημείωση των πρόοδου όσον αφορά του περιβάλλοντος και θα πρέπει να δούμε πρώτα πρώτα τι γίνεται όσον αφορά τη δική μας βιομηχανική βάση. Όμως, Εάν οι αποφάσει μας αφήνουν περιθώριο για τέτοιες διατυπώσεις, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακριβώ αυτό το είπε η κυρία Μέρκελ στην ε, ομιλία της στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιμάνης και ο κύριο Κουάντρας. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα ευχαριστίες στην κυρία Χίμνερ για τη δουλειά της. Σύμφωνα με το όσο προτείνει, επιβάλλεται να προβληματιστούμε. Για το τι γίνεται με τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα που συχνώνονται σε ΙΠΑ Ευρώπη, αλλά αυξάνονται στην υπόλοιπο κόσμο. Αν μην ξεχνούμε δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί μόνο το 11% των εκπομπών του διοξείδου των ανθρώπου παγκοσμίω στο μέλλον. Πρόκειται να κατεβάσουν εκπομπές από αυτή τη συμμετοχή μας. Βέβαια, ο πληθυσμό αυξάνεται. Και άρα και η κατανάλωση ενεργείας αυξάνεται. Έχουμε λοιπόν αυτήν την αντίθεση μεταξύ των προσπαθειών που καταβάλλονται στην Ευρώπη και από την άλλη μεριά την αύξηση των εκπομπών παγκοσμίω. σε αυτό το πλαίσιο επομένω δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Χίμπνερ αλλά και με τον κύριο Σιμάνσκι. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το τι διαβήματα κάνει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές. Να δούμε και τι γίνεται με την βιομηχανικότητα, μια προσπαθούμε να κάνουμε κάποιο είδου ε, έγκαιρα βήματα και να προσπαθήσουμε να έχουμε βιώσιμη οικονομία. Επίσης, θα πρέπει αποφασιστικά να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους άλλους, να συντονιστούν με τις παγκόσμιες προσπάθειες για να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή. Επίσης, θα πρέπει μεγάλη προσοχή να σταματήσουμε τον αθήμενο ανταγωνισμό η βάρα της βιομηχανίας μας. Πάντως, είναι σαφές ότι φέτος η διάσκεψη στην Βαρσοβία θα πρέπει να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους από ό,τι στο παρελθόν. Στην Τόχα συνειδητοποιήθηκε το πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ενιαία φωνή Ευρώπη. αυτό και ήταν σημαντικό το ότι είχαμε αυτή τη συμφωνία πριν την διάσκεψη. το πολιτικό φάσμα από όλες τις χώρες. Οπότε και έτσι εξοικονομούμε χρόνο προσπάθεια για όταν έρθει η ώρα της συνάντησης. Σύμφωνα με την κυρία Χίπνερ για το πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Αυτός είναι ο τρόπος να μειωθούν οι εκπομπές και ορθά θεωρεί, κύριε Χίμπνερ, ότι είναι προτεραιότητα η, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Και αυτό αποτυπώνεται στην εκθέσή της. Η πρόεδρος, η κυρία Χολ. Μαδάμ Καρβάλιο. Δεν παρίσταται και έλαβε το λόγο κυρία Καρβάλιο. Thank you, Chair. Uh, I Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι εις θέση να έχει το ανταγωνιστικό εκτίμα. επί τη βάση της πλατφόρμας του Ντέρμπαν. Άρα, να καταλαβαίνουμε το ότι η ΚΟΠ επανέρχεται. Άρα και εμείς στο ψήφισμά μας να Πού είμαστε στην Επιτροπή ότι πρέπει να λάβει υπόψη αυτέ τις βασικές μας ε, προτάσει, ε, πιστεύω, αρχέ. Πρώτα πρώτα, αυτή η μέτρο συμφωνία δεν θα πρέπει να χωρίσει τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Ακριβώ όπω έκανε το πρωτοκόλλο του Κιώτο, που χώρισε τον κόσμο σε βιομηχανικέ χώρε και σε αντισώμενε χώρε. Δηλαδή, οι στόχοι προ επίτευξη ε, βρίσκονται και απόκεινται από τις ε, βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες και επομένως θα πρέπει να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας, να έχουμε ας πούμε κάποια κριτήρια όπως με το ΑΕΠ κατά κεφαλή, επίπεδο εκπομπών, τεχνολογίας, τέτοια κριτήρια και δείκτες που να είναι εύληπτη. Επίσης, έχουμε κάποιους στόχους και από συγκεκριμένους κλάδους της ε, βιομηχανίας. Και μπορούμε να συνδυάσουμε ένα τομέα με κάποιον άλλο. Ή τόσο να συνδυάσουμε ένα τομέα με κάποιον στόχο, τομιακό, ας πούμε. Οπότε έτσι να ε, μην έχουμε διαρροές από τομείς Βιομηχανική παραγωγή που χρειάζεται από ένταση. Και να έχουμε επίση και αυτέ τις πρωτοβουλίε, πρωτοβουλίε από τη βάση, όπω πρωτοβουλίες των πόλεων. Επίσης ο μηχανισμός της αγοράς θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, να βελτιωθεί, ακριβώ όπω το TTS και το CDM Επίση θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει, αλλά θα πρέπει να απλουστευτεί. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών και να αποτελούν πιο ενέργειε. Επίση, να υπάρξει συνεργασία όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη και ο πρόεδρο Ομπάμα αναφέρθηκε στην αγορά τη καθαρή τεχνολογία που θέλει να συγκροτήσει στη συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή, μπορούμε να τη βάλουμε στο κείμενό μας. Όλο αυτό το κείμενο που σας ανέπτυξα τώρα θα το στείλω σαν σημείωμα στην εισηγήτρια. Πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που προηγήθηκαν. Εγώ είμαι ιδιαίτερα επιφυληκτικός για τη δυνατότητα να συνάψουμε διεθνείς συμφωνίες. Ως τώρα δεν έχει δοθεί καμία απόκριση στη δήλωση του Μπαλή για την common but differentiated ευθύνη, για την κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη. Θεωρώ ότι αυτό είναι κεντρικής σημασίας, εάν επιδιώκουμε διεθνή συμφωνία. Μία συμφωνία που δεν θα είναι διεθνής δεν θα έχει και νόημα. Με το Κιώτο προκρίναμε την επιλογή ενός μηχανισμού της αγοράς ένας μηχανισμός όμως που βασίζεται στην αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει αν το 50% των δικαιωμάτων εκπομπών δεν διανέμονται δωρεάν. Και εάν ε, υπάρξουν ε, επεισόδια όπως αυτά που συνέβησαν με το clouding. Αλλά αυτό ήταν μια παρέμβαση στο μηχανισμό αγοράς και ελπίζουμε τέτοια επεισόδια να είναι σπάνια και αν γίνεται και μοναδικά. Το Κιώτο καθόριζε την διάκριση μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών, όπω μόλι τώρα επενθυμίστηκε. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά, διότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα, ε, πρέπει να επιδιώξουμε μια διαφορετική τελείω πρόταση, βασισμένη στην ισοτιμία, την δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά το βιώσιμο επίπεδο των ε, δικαιωμάτων εκπομπών ε, αερίου του θερμοκηπίου. Αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να μοιραστούν ισότιμα και δωρεάν σε όλους τους κατοίκους αυτού του πλανήτη, σε όλους τους ανθρώπους. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να ε, εκπέμπονται με αντίτιμο, βάσει αντίτιμο. Αυτό λέει και η δήλωση του Μπαλή. Χρειάζεται λοιπόν τόλμη και πυγμή, ιδάλλως ας τα αφήσουμε να χαθεί. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρίσταται. Υπάρχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή καλωσορίζει την συζήτηση που έγινε από τους βουλευτές για την προετοιμασία της διάσκεψης των μερών COP19. Ακούστηκαν πολλές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης το θέμα των εκπομπών που αυξάνονται, κλιματικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, οι τάσει ενεργειακή κατανάλωσης, ο ρόλος της ενεργειακής αποδοτικότητας, της βιομηχανίας, οι ανάγκες των καταναλωτών, η ανταγωνιστικότητα, οι τεχνολογικές λύσεις, οι βασικές αρχές όπως η συμμετοχή όλων, ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν κόσμο διερευμένο στα δύο μέσα σε μια συμφωνία τις αντιδράσεις, τις πρώτες προτάσεις, τα προβλεπόμενα ωφέλη, τα βασικά στοιχεία των προηγούμενων συμφωνιών, του πρωτοκόλλου του πρώτου και το καθεξής και το καθεξής. Όπως ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη νέα συμφωνία που πρόκειται να εγκριθεί το 2015 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2020 και έχουν ξεκινήσει ήδη οι προετοιμασίες. Ήδη στη Βόνη ε, είχαμε κάποια ενθαρρυντικά δείγματα για τα νέα προβλεπόμενα στοιχεία της ε, επόμενης συμφωνίας. Θα πρέπει να είναι νομικώς δεσμευτική και να έχει παγκόσμια εμβέλεια, να είναι εφαρμοστέα δηλαδή σε όλους, με έναν κοινό στόχο ε, μείωση και αναχέτησης της αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασία κατά δύο βαθμούς Κελσίου. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε στο τέλος του 2015. Σημειώνω αυτά που είπε η συγγήτρια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να πολεμήσει μόνη ε, σε ένα διεθνή ωκεανό δηλαδή να, ε, να πελαγοδρομεί μόνη, αλλά θα πρέπει οι μεγάλες οικονομίες παγκοσμίω να συμμετάσχουν βάσει των εθαρρυντικών μηνυμάτων που έχουμε από τις ΗΠΑ, από την Κορέα, από το Μεξικό, από αρκετούς άλλους σημαντικούς φορείς όπως η Κίνα Μπορεί και να γίνει αυτό. Ε, το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων κομπών ε, του αερίου θερμοκηπίου στην Κίνα και στι ΗΠΑ είναι ήδη κάποια μηνύματα. Είναι ενθαρρυντικά, αλλά θα χρειαστεί ακόμα πολλή δουλειά. Και την έχουμε μπροστά μα τη δουλειά αυτή. Οι πρόσφατε συζητήσει στη Βόνη έδειξαν ότι του χρόνου, το 2014, θα είναι καθοριστικό έτο. Θα είναι το έτο των φιλοδοξιών. Τότε περιμένουμε και ελπίζουμε να έχουμε πλέον συγκεκριμένε προτεραιότητε με φιλόδοξε δεσμεύσει φιλόδοξες υποσχέσεις, καθώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της χρηματοδότησης σε αυτή τη φάση. Επίσης ένα καθοριστικό ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί στη Βαρσοβία με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εν το 2015 είναι η σταδιακή προσέγγιση, βήμα προς βήμα. Θα πρέπει να καταρτήσουμε και το ρόλο των σχέσεων συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, του αποτυπώματος άνθρακα και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Και Τέλος, εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να θυμόμαστε τη δεύτερη φάση δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιώτο που έπρεπε να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Τροπή και τα υποβάλλει σύντομα πρόταση για το θέμα αυτό και ελπίζουμε στη στήριξή σας και εδώ, όπως και στο παρελθόν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την ολοκλήρωση της συζήτησης. Ο λόγος του συνάδελφου Χίμπνερ. Τρία λεπτά. Γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να παραδεχτώ ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους έθιξαν ζητήματα τα οποία σημειώνω Τίποτε δεν θα παραμελήσω και όλα θα τα εξετάσω ε, για να απαντήσω στο συνάδελφο Σιμάνσκι. Αφού προσπαθήσαμε να μην ε, ανατρέξουμε σε έγγραφα που δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένα και δεν συνέβαλαν στον επιτελεστή πρόοδος, προφανώς όπου πειραθήκαμε η πρόταση να προτείνει και μία διάγνωση αλλά και μία διέξοδο από τα προβλήματα. Βεβαίω και αναμένουμε να προταθούν συγκεκριμένε χειροπιαστέ λύσει. Δεν υπονοώ ότι κάποιοι προσπαθούν να μα παγιδέψουν ή ότι είμαστε απομονωμένοι. Προσπαθούμε όμως να αναλύσουμε πώς έχουν τα πράγματα γύρω μας και θα θέλαμε όλοι να αγωνιστούμε από κοινού. Να αγωνιστούμε από κοινού για την επιτυχία της παγκόσμιας βιομηχανίας. Προφανώς υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά ακόμα και σε μια ανταγωνιστική βιομηχανία, εφόσον τεθούν σωστά οι προδιαγραφές και τα πρότυπα, μπορούν όλοι να έχουν ίση συμμετοχή. Και παρά την... Ε, αντί μάλλον να ψάχνουμε να εντοπίσουμε εχθρούς, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε όλοι αναγκασμένοι να συνεργαστούμε. Είναι πολύ ωραία το παράδειγμα της κυρίας Μέρκελ, αλλά θα πρέπει να δούμε πού μπορεί να επιτελεστεί πρόοδος. Ε, η ανταγωνιστικότητα λοιπόν της ευρωπαϊκής μηχανίας είναι κάτι που όλοι το επιθυμούμε. Μην ξεχνάμε τους κλιματικούς στόχους από τη μία, αλλά από την άλλη να έχουμε και το βλέμμα στραμμένο στον ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο συνάδελφος η Ευρώπη να μιλάμε ενιαία φωνή και όχι να υπάρχουν αναταράξεις. Ε, το Συμβούλιο να λέει το ένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κάτι τρίτο. Πρέπει να έχουμε μια κοινή τοποθέτηση, μια κοινή στάση. Και βεβαίως θα λάβει υπόψη σοβαρά τις προτάσεις της συναδέλφου Καρβάλιου, ώστε να προσθεθούν κάποια στοιχεία. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πρόντι και να πω ότι δεν πιστεύω τόσο στο πρωτόκολλο του Κιώτο, ούτε εγώ ίδια. Δεν είναι η μόνη καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Με τις διατάξεις που τώρα έχουμε στα χέρια μας, τελικά δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας, αλλά να είμαστε και στραμμένοι προς το μέλλον. Θα πρέπει να ξέρουμε κάτι που να είναι εύληπτο για όλους και αποδεκτό από όλους. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ και ξεκινάμε αμέσως τη συζήτηση στην κυρία Τζαβέλα για την ανάπτυξη ποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Έχουμε στη διάθεσή μας έχουμε στη διάθεσή μας για τη συζήτηση περίπου 20 λεπτά. 5-7 λεπτά, κυρία Τζαβέλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το πλαίσιο που μας δίνει η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές υποδομές έτσι θα διευκολυνθούν οι νεοεισερχόμενοι σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά και θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Επί του παρόντος είναι δύσκολο για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα οχήματα να ανταγωνιστούν στην εσωτερική αγορά και να αποτελέσουν ένα σημαντικό κομμάτι της. Για παράδειγμα, τα οχήματα που δεν χρησιμοποιούν προϊόντα πετρελαίου έχουν δυσκολίες να πουληθούν στην εσωτερική αγορά διότι οι επιλογές του ανεφοδιασμού ή επαναφόρτηση δεν είναι άμεσα διαθέσιμες τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν σε γενικές γραμμές καλωσορίζω αυτή την πρόταση της Επιτροπής και τις προσπάθειες για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων που στοχεύουν στη σταθερή μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από το πετρέλαιο. Πιστεύω ότι οι επενδύσεις θα πρέπει πρωτίστως να οδηγηθούν σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς και θα πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια τεχνολογικά ουδέτερη βάση. Επιπλέον πιστεύω ακράδαντα ότι τα κατάλληλα κεφάλαια για την έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να διατεθούν από την Ένωση προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αγορά και να επιταχυνθεί η ετοιμότητά τους για υλοποίηση. Έχω καταθέσει σχετική τροπολογία επ' αυτού. Επίσης, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τυποποίηση είναι κρίσιμη σημασίας, δεδομένης της μεγάλης διασυνοριακής διάστασης της παρούσας οδηγίας. Δεν θα έπρεπε αυτή η οδηγία να είναι το πεδίο μάχης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, για το τι τύπου πρίζα θα χρησιμοποιούμε σε όλη την Ευρώπη πάνω σε αυτό το θέμα μέσα από συγκεκριμένη τροπολογία προσπάθησα να βρω μια συμβιβαστική λύση σε αυτή τη διαμάχη και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την τροπολογία. Υπάρχει και η γεωπολιτική σημασία αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις στη ΣΥΠΑ, στις οποίες η Επιτροπή ίσως δεν πρόλαβε να εστιάσει ή να δώσει την απαιτούμενη έμφαση. Αν φτάσουμε σε σημείο που από ό,τι διαφαίνεται εκεί ε, οδηγούμαστε, σε τρία-τέσσερα χρόνια να έχουμε εξαγωγές και πετρελαίου από τις Ηνωμένε Πολιτείε, πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Το πετρέλαιο δεν φαίνεται να φεύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή μας. Από την άλλη πλευρά, η φθηνή παραγωγή του φυσικού αερίου στη ΣΥΠΑ οδηγεί σε περισσότερο φυσικό αέριο που θα είναι διαθέσιμο στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΑ, η Κίνα αλλά και η Ευρώπη μπορούν να αναπτύξουν νέα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Μια τέτοια μεταφορά εναλλακτικών ορυκτών καυσίμων δημιουργεί κίνητρα για την μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, στα αυτοκίνητα και στους τόλους μεταφορών. Επιπρόσθετα η προοπτική των home refueling kits είναι ενδεχομένως κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά για τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Αυτά τα kits είναι πιθανόν να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα το 2017-2018. Θα έπρεπε και η Ευρώπη να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό στην πρόταση της Επιτροπής και σκοπεύω να καταθέσω τροπολογίες πάνω σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να ζητήσω τη στήριξή σας. Εφόσον μιλάμε για κάτι καινούριο, είμαι διατεθειμένη να δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ναι μεν πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστές η Ένωση το καλύτερο που έχει να κάνει σε τέτοιες προσπάθειες είναι να προσφέρει μέσω χρηματοδότησης για την έρευνα, για την έρευνα και να προβεί σε ενέργειες τυποποίησης που μπορούν να διευκολύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Προσδοκώ να ακούσω τις γνώμες πάνω σε αυτό το, θέμα, τις γνώμες όλων σας και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζαβέλα. Και τώρα το λόγο στους και οδησηγητές σε τρία λεπτό καθένα σε Μπρετζίνα, ο πρώτος. Ευχαριστούμε κύριο Μπρετζίνα. Όσον αφορά τώρα την εναλλακτική παροχή καυσίμων, νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολύ καλέ ιδέε για από αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Τζαβέλα. Εδώ πέρα υπάρχουν προτάσει για διάφορε πρωτοβουλίε. Για ε, το, το φυσικό αέριο, το υδρογόνο, Όλα αυτά ως καύσιμα, όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιχαραγωθούν και να οριστούν και θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες ε, υποδομές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ε, ποια θα είναι η απόσταση μεταξύ των διαφορετικών σημείων ε, προμήθειας των καυσίμων και θα πρέπει επίσης να δούμε και πώς θα ρυθμίσουμε τα της παραγωγής και διάθεσης αυτών των διαφορετικών καυσίμων. Θα πρέπει να γίνει επομένως μια ευρωπαϊκή ή παγκόσμια προσπάθεια εναρμόνισης και πρόκειται για θέμα και διασυνοριακό. Τέλος πάντων θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ανεφοδιασμού πάντως στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη τα οποία θα εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο δίκτυο θα πρέπει να έχουν λίγο αυτά τα κράτη-μέλη ένα ε, περιθώριο ελιγμών τους ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν στην επιτευξή των στόχων όπως αυτοί έχουν οριστεί. Διαβάζω τις τροπολογίες, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλό το κείμενο, αλλά όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να αναφέρουμε διαφορετικούς τρόπους ε, ανεφοδιασμού. Ας πούμε, για τις επαγωγής υπάρχει ένας τρόπος που δεν αναφέρεται εδώ, τρόπος ανεφοδιασμού. Τόσο τον ευχαριστώ την κυρία Τζαβέλα και τους άλλους και οδησίγητες. Σας ευχαριστώ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Λάγκεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως ε, όταν ε, καταρτίζουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με πολλά χρήματα, θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον είναι σωστές οι προδιαγραφές. Και έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, δεν κατάλαβα καλά κατά πόσον το κριτήριο για την επιλογή χώρων ε, εφοδιασμού για τις ε, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ε, κατά πόσον η απόσταση μεταξύ τους είναι σωστή. Δηλαδή το να πούμε ανά 150 ή ανά 200 χιλιόμετρα, αυτό ε, ενδεχομένως σημαίνει ότι τοποθετείται χώρος ε, ανεφοδιασμού όπου ένα αυτοκίνητο πάει από το Ρις στη Στοκχόλμη αλλά ας πούμε στο Παρίσι θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότεροι σταθμοί ανεφοδιασμού γιατί εκεί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πούμε έτσι άκαμπτα ότι το κριτήριο για τους σταθμούς αναφοδιασμού είναι η απόσταση μεταξύ τους αν δεν έχει κανείς προηγουμένως μελετήσει τη ζήτηση. Ε, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω ε, σε σχέση με τις προδιαγραφές για τις μπρίζες ε, και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Στα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα έχουμε δύο είδη ανεφοδιασμού. Έχουμε καταρχήν τον απλό κανονικό ανεφοδιασμό με το σύστημα ACAC που συνδέεται με την πρίζα υπαριθμών 2 και συμφωνήσαμε από αυτού. Όμως κυρίες και κύριοι αυτός ο ανεφοδιασμός ε, διαρκεί 8 ώρες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει νόημα να ε, κατασκευάσουμε σταθμούς ανεφοδιασμού που θα είναι μακριά από το σπίτι ή από το χώρο εργασίας ενός ανθρώπου. Δεν θα περιμένει κανείς 8 ώρες να ανεφοδιαστεί το αυτοκίνητο. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει να συνδυάσουμε ε, τους, ε, τις μπρίζες να είναι συνδυασμένο το σύστημα AC με το DC να είναι σαφές αυτό ε, σχετικά με τις προδιαγραφές έτσι ώστε και η ευρωπαϊκή βιομηχανία να γνωρίζει τι είδου ε, μπρίζες και υποδοχές πρέπει να κατασκευαστούν για να μην γίνουν λάθη. Τώρα, άλλο ερώτημα έχει σχέση με τη χρηματοδότηση. Νομίζω και αυτό ε, πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Αν θέλουμε να φτιάξουμε μια πραγματική υποδομή, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτούς που αργότερα θα πουλάνε τα καύσιμα αυτά έτσι ώστε να ε, συμπεριλάβουμε και το στοιχείο της οικονομικής απόδοσης. Ε, πιο σημαντικό είναι αυτό από το να κατασκευάσουμε ένα σωρό σταθμούς που ενδεχομένως μετά να είναι άχρηστοι. Γι' αυτό λοιπόν να σκεφτούμε τα κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν ε, πραγματικά αυτά να εξυπηρετήσουν τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης. Αουλ. Κύριε να ευχαριστήσω την ε, εισηγητρία για Πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί τη και είναι πάρα πολύ θετική πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής γιατί εξαρτώμαστε τόσο πολύ από το πετρέλαιο. 94% είναι η εξάρτησή μα. Και σκεφτείτε πώς κοστίζει αυτό και πόση λίγη ασφάλεια ανεφοδιασμού έχουμε. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, υπερθέρμανση του πλανήτη, θα πρέπει τουλάχιστον 60% μέχρι το 2050 να έχει σταματήσει η εξάρτησή μας από ε, ενέργεια που εκπέμπει διοξίδιο. Άρα, θα πρέπει να έχουμε κατάλληλη υποδομή, ώστε να απομακρυνθούμε από αυτές τις μορφές ενέργειας που μας οδηγούν στην εξάρτηση. Θα πρέπει επίσης να έχουμε και να εφαρμόσουμε κάποια πρότυπα για αυτή την υποδομή. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει κάποια εναρμόνιση και εναρμοσμένη ρύθμιση μάλλον για τα σημεία εφοδιασμού γιατί θέλουμε και εδώ είναι αγορές θα πρέπει τώρα να δώσουμε μεγαλύτερη προθεσμία, μικρότερη προθεσμία για τις ορισμένες ε, περιοχές. Υπάρχει πρόβλημα. σε σχέση με τα πρώτα που προτείνονται στο τρίτο παράδειγμα, Επομένω, θα πρέπει εκείνε οι περιοχέ που έχουν το πρόβλημα να έχουν λίγο περισσότερο χρονικό περιθώριο για να μπορούν να προσχωρήσουν στο νέο πρότυπο. Τώρα για την ανάλυση κόστου ωφέλου. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το ζητήσουμε αυτό να το κάνει το κάθε κράτο μέλο. Θα έπρεπε κανεί να κάτσει να δει πόσο κοστίζει Σήμερα η κατάσταση με το πετρέλαιο για τις εκπομπές του δεξιδίου. Είναι αδύνατον τα κρατημέλη να κάνουν κάτι τέτοιο, αν τους το ζητήσουν. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε τον πηγή ψηλά και αν δεν μπορούν τα κρατημέλη μας το πούν. Για το ευρωγόνο το στο άρθρο 5 λέει ότι θα πρέπει η υποδομή να αφορά όλη την επικράτεια. Μα σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα ή η Βρετανία που έχουμε τόσα νησιά δεν είναι τόσο ρεαλιστικό αυτό. Και στο πρέπει να λέμε ότι θα πρέπει σε όλη την επικράτεια του υπηρετικού τμήματος τη χώρα να υπάρχουν αυτά τα σημεία εφοδιασμού. Άρθρο 4, παραγωγός 6, κάτι λέει για έξυπνα ε, δεν είμαι σίγουρη ότι χρειάζεται. αυτό αυτού τα ρολόγια μέτρηση της χωρίς χρειάζεται όταν κάποιος έχει στο σπίτι του ανεφοδιασμό. Α πούμε σε ένα σημείο δημόσιο, κάνει ένα στα ψώνια του και την ώρα που τα κάνει έχει βάλει την πρίζα και φορτίζει το αυτοκίνητο. Επίσης, στο γήμα της πρότασης αναφέρονται διάφοροι τρόποι ανεφοδιασμού, ούτως ώστε να καλύψουμε και τις εξελίξεις τεχνολογίας. Άρθρο 4, παραγραφός 8. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί πάροχοι. Είναι θέμα ανταγωνισμού, τέλος. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να επιμείνουμε στο να υπάρχει προτυποποίηση όσον αφορά το, το σωλήναν εφοδιασμό. Δεν έχει ο καθένας το, το, το σωλήνα που θέλει. Να ταιριάζουν επομένως σε κάθε μόνο εφοδιασμό, σε με το, το, το, την υποδοχή του οχήματος. Ο κύριος ε, Τοζανόφσκι. Και εγώ ε, θα ήθελα να ε, πω ότι χαίρομαι για αυτό το κίνημα και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Όπως το επηρεάζει συνάδελφος, είναι μια δύσκολη συγκυρία αυτή για να το συζητήσουμε, γιατί ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι ποια τεχνολογία τελικά πρόκειται να επικρατήσει. Άρα θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά το πώς θα ορίσουμε τα αναγκαία διοικητικά μέτρα. Ακόμα είναι νωρίς. Δεν έχει επικρατήσει καμία ιδέα. Θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη για το κείμενο και όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά τα καύσιμα. Όπως είπε ο κύριος Λάγκε, και εγώ απορώ πώς θα ορίσουμε και θα καθορίσουμε την απόσταση μεταξύ των σταθμών εφοδιασμού γιατί έχουμε μεγάλη ποικιλία στην γεωγραφία, στη μορφολογία κάθε χώρας. Ιδίω για τα ιδιωτικά σημαίνει φωτισμό. Πώς θα στηθούν αυτά, μια που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Τώρα όσον αφορά τους σωλήνες ε, σύνδεσης, τον τρόπο σύνδεσης του οχήματος, με, ε, στο σήμερα εφοδιασμό. Να, θυμάστε πώς έχει κατάσταση με τα κινητά και τα τροφοδοτικά τους. Τελικά όμως, από το χάος το αρχικό κάπου σταθεροποιήθηκε η κατάσταση. Μέχρι σήμερα έχουμε περιορισμό, ας πούμε, από την μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να είναι φορτισμένη. Ε, αυτό είναι ένας περιορισμός, είναι ένας φραγμός. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τη δυνατότητα της κάθε μπαταρίας σε σχέση με τον καθορισμό της απόστασης του κάθε σημείου εφοδιασμού. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Θα πρέπει να ξανοιχτούμε στα βαθιά, να προβληματιστούμε και να καταλήξουμε σε κάποια προτυποποίηση. Να καθορίσουμε και τα σημεία φοβιασμού, τι θα τα διέπει, αλλά μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τα κρατημέλη, γιατί οι καταστάσεις διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος στο άλλο. Επίσης η αγορά ακόμα δεν έχει δείξει. Τι δρόμο πρέπει να πάρουμε. Τόσο νομίζω ξεπέρασα το όριο αγόρευση, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο μου, τον Ζανόφσκι σε για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που με απασχολούν και με ανησυχούν. Αυτά που προτείνονται είναι πολύ ακριβά, πολύ δαπανηρά. Ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη η γεωγραφική θέση ορισμένων κρατών μελών αλλά και η τεχνολογική τους εξέλιξη. Δεν έχουμε σε όλα τα κρατη την ίδια τεχνολογική εξέλιξη. Υπάρχουν κάποια κράτη που είναι ε, πιο φτωχά, στο πούμε απλά, στα ανατολικά της Ευρώπης και αυτό θα αποτελούσε επιβάρυνση στα δημοσιονομικά τους. Ε, με την πρόταση αυτή η ε, Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, κάποιες προχωρημένες τεχνολογίες αλλά αυτές δεν είναι ακόμα έτοιμες για την αγορά και αυτό με απασχολεί. Θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω και τις δαπάνες. Η Κομισιόν έχει κάνει μία ε, αξιολόγηση, αλλά δεν είναι σωστή αυτή η αξιολόγηση. Είναι κάτω από το προβλεπόμενο. Γίνεται λόγος ή πρέπει μάλλον να γίνει λόγος για σταθμούς εφοδιασμού, ε, στους σταθμούς αυτούς ε, να υπάρξει σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αφορούν στην υποδομή και το οικονομικό βάρος. Ποιος θα το επιφορτιστεί, ο ιδιωτικός τομέας ή μήπως και οι καταναλωτές. Αυτοί θα πληρώσουν το Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στα φτωχά κράτη-μέλη ε, που και οι πολίτες εκεί έχουν περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Ε, κάτι άλλο, ίσως ε, και οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και αυτές να μην είναι ασφαλείς, γιατί μιλάμε για αγορές που ενδεχομένως να μην τύχουν πλήρους εκμετάλλευσης. Μιλάμε δηλαδή εδώ τελικά για τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα οριμάσει. Πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο να οριμάσουν. Για όλους αυτούς τους λόγους τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πρόωροι αυτή η χρήση. Και κάτι άλλο, όσον αφορά ε, τα εναλλακτικά καύσιμα, εάν αυτά φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα παρουσιακά, παραδοσιακά, ε, δεν θα υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Το δίζελ, ας πούμε, φορολογείται κατά 40% λιγότερο από το πετρέλαιο. Μην το ξεχνάτε. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, σίγουρα αυτά θα ε, περιοριστούν, αλλά μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή ενέργειας, αυτό θα μπορούσε να γίνεται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων και αυτή πάλι θα οδηγήσει σε εκπομπή διοξιδίων του άνθρακα. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Επειδή ε, μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από πηγές ενέργειας, αυτή η πρόταση Κομισιόν καταρχήν είναι ευπρόσδεκτη. Βεβαίως ένα από τα βασικά εμπόδια χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι η ηλεκτρική ενέργεια και βεβαίως και η ύπαρξη σωστής υποδομής αυτές οι πηγές ενέργειας πρέπει να δημιουργούνται με αποθήκευση, ενδεχομένως να υπάρχει μεταφορά και διανομή ενέργειας. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει και η κυρία Τζαβέλα, οι σταθμοί εφοδιασμού ακόμα δεν υπάρχουν. Παρόλα αυτά, η κυρία Τζαβέλα υπογραμμίζει επίσης ότι οφείλουμε να προσέξουμε και το κόστος παραγωγής ε, εναλλακτικών ε, καψίμων ε, που είναι πολύ πιο μεγάλο από τα παραδοσιακά καύσιμα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε τη σχέση κόστους-οφέλους σε αυτές τις επενδύσεις και να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που συνδέονται με όλα αυτά. Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι πραγματικά εναλλακτικά εάν αυξηθεί και το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προς το παρόν αυτό δημιουργεί πρόβλημα τουλάχιστον στις μεγάλες αποστάσεις. <clears throat> Σημερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες της κυρίας Τζαβέλα σχετικά με την οριμότητα του αυτοκίνητου κινούμενου με υδρογόνο και τους ε, κινδύνους ε, που υπάρχουν στο να επενδύσει κανείς σε τέτοιο είδους ε, υποδομή όταν αυτή δεν έχει τελειοποιηθεί. Κρίμα που δεν είναι εδώ ο κύριος Πρόντι γιατί είμαι σίγουρος ότι εκείνος θα μας παρουσίαζε μια πολύ πιο αισιόδοξη προοπτική. Τέλος να πω Ελπίζω η πρόταση αυτή μαζί με την άλλη που συζητάμε για τα βιοκαύσιμα και οι δύο θα συμβάλλουν στο να περιορίσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση και να γίνουν οι μεταφορές μας πιο πράσινες. Όμως ε, ποτέ δεν ε, πρέπει να ε, αγνοούμε το ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Πολύ ωραία λέει πρόεδρος, πρώτα η Κομισιόν ε, και μετά η κυρία Τζαβέλα θα λάβουν ε, το λόγο η Κομισιόν, ε, δύο λεπτά παρακαλώ, γιατί έχουμε καθυστερήσει για την επόμενη σύντηση με την Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τζαβέλα για το σχέδιο της γνωμοδότησής της, που αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξουν κίνητρα και να σταλούν μηνύματα ε, στην αναγκαιότητα δημιουργίας υποδομής έτσι ώστε να διευκολυνθεί η θέση σε αγορά των καθαρών αυτοκινήτων. Επίσης, ε, πολλοί συνάδελφοι έχουν δίκιο, η Ευρώπη εισάγει ενέργεια για την κινητικότητά της, άρα δηλαδή είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική αγορά. Αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα αυτή τη στιγμή δεν εξαπλώνονται λόγω του ότι είναι δαπανηρά και δεν υπάρχει και η υποδομή για τον εφοδιασμό. Ε, διασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει έναν, τουλάχιστον έναν ελάχιστο αριθμό σταθμών εφοδιασμού μπορούμε με τον τρόπο αυτό να σπάσουμε το φαύλο κύκλο όπου ε, δεν θα ε, υπάρχει απαράδεκτη επιβάρυνση για κανένα. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία, εν πάση περιπτώσει, που προκαλεί την ε, προσφέρει μάλλον δυνατότητες για επενδύσεις στην αγορά. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο το να εισαχθούν εναλλακτικά κάψιμα για να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως είναι έλλειψη εμπιστοσύνη από πλευράς ε, κατανοητή και έλλειψη τεχνολογικής πρόοδου. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υφίστανται, ε, η άποψη τεχνολογικά καθαρά είναι ουδέτερη. Έχουμε λοιπόν και δεσμευτικούς ε, στόχους ε, ε, για τους σταθμούς εφοδιασμού. Αυτά έχουν σχέση και με την οριμότητα των κρατών μελών. Όπως είπε και η συγγήτρια, αυτό που έχει σημασία είναι η ευρωπαϊκή αγορά να παραμείνει στην πρώτη γραμμή γιατί σε σύγκριση με τις Ηνωμένες και την Ιαπωνία έχουμε ήδη καθυστερήσει. Η Νίκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ε, ορθολογικές παρατηρήσεις που κάνανε. Έχω σημειώσει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς και προσβλέπω σε μια παραγωγική και αποτελεσματική συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, veramente bravissima. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήσασταν λακωνικότατοι. Ε, το ε, Σεπτέμβρη έχουμε την καταληκτική ημερομιλία για την κατάθεση των ε, τροπολογιών. Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είπαμε στην Επίτροπο να έρθει λίγο αργότερα. Η κυρία Τράουτμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κάποιες σκέψεις. Να μην επισέλθουμε σήμερα στις ε, λεπτομέρειες μια που πιεζόμαστε χρονικά. Και θα πρέπει σε λίγο να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα την κυρία Κρούς. Να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους για τις ε, συμβολές τους, προφορικές και έγγραφες και να σας πω ότι ο στόχος εδώ είναι να αναλύσουμε αυτήν την οδηγία πλαίσιο σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες, ότι θα ισχύσει, ότι ισχύει μάλλον μόλις από τον Ιανουάριο στο τέσσερα του κρατημέλη. Έχουμε αυτή την νομοθετική πρόταση του 2007 και επίσης ε, ε, ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσει το 2009 για να καλύψουμε τις πολυπλοκότητες του αυτού του πακέτου επικοινωνιών και να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Και θα πρέπει πρώτα πρώτα να σας διφωνήσω κάτι. Ο στόχος μου δεν είναι με κάθε τίμημα να προστατεύσουμε το κράτος. Δεν θέλω να θεωρήσω ε, ότι, είναι το ιερά και τα όσια δηλαδή, γιατί έχουμε και αυτόν τον τρόπο κλείσει εκείνο το συμβασμό με το Συμβούλιο και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει ε, κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που είναι προσαρμοσμένο στην εξέλιξη της τεχνολογίας και θα πρέπει αυτό να ε, συνδέεται με την κατάσταση της αγοράς. Τώρα, πλευράς μεθοδολογίας. Ακόμα δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να κρίνουμε αν πετύχαμε ή αν αποτύχαμε. ούτε να μιλάμε για βραχυπρόθεσμη αναθεώρηση. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η αξιολόγηση. Να δούμε τι έχει αποδώσει λόγω του πακέτου επικοινωνιών και τι πρέπει να βελτιωθεί. Τι έχει αξιοποιηθεί ή όχι. Θα δούμε επομένω ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να τα ξαναδούμε τα ζητήματα αυτά εις την επόμενη θητεία. Γι' αυτό και εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το κείμενο άρθρο-άρθρο και επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια μελέτη εις βάθος. Γιατί? Θα πρέπει ο νομοθέτης να μην παραβλάψει το προβλέψουμε τον εξελίξουμε σε αυτόν τον κλάδο, γιατί μόνο έτσι γίνονται κατάλληλε επενδύσει. Έτσι θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Και να, πρέπει να συμφωνήσει τελικά το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο για αυτή την νομοθετική πρόταση. Ο στόχος αυτής της έκθεσης της πρωτοβουλίας είναι να δούμε στη συνέχεια σε τι θα πρέπει να προβληματιστούμε στη δεύτερη φάση να δούμε τι ισχύει στην αγορά, να δούμε αν θα πρέπει να γίνει ε, κανονιστική ρύθμιση εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων και πρόκειται εδώ για μια ρύθμιση που θα έχει σημαντικές οικονομικές ε, επιπτώσεις όπως με το άρθρο 7 7. Και ξαναλέω θα πρέπει να είναι τέτοιο το νομοθετικό πλαίσιο που να ε, ελκύει τις ε, επενδύσεις. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα του κλάδου. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια που θα φέρει την αναγκαία ασφάλεια, ούτως ώστε να είναι, κατα... να είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής. Από τις αντίσεις που είχα κατάλαβα ότι το σημερινό πλαίσιο δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη πολιτική βούληση των ε, καταμελών. Και γι' αυτό τίθεται το θέμα του πόσο εύστοχη είναι η νέα νομοθετική πρόταση. Και επίσης θα πρέπει να ε, δούμε τι λέει το άρθρο 15 παραγραφός 4 εκεί που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει τις ε, διεθνείς αγορές ε, επίσης το μηχανισμός της κατανομής του ρίσκου, του κινδύνου και επομένως πρόκειται για κάποιες προσθέσεις, προσθήκες ή τροπολογίες ή ε, τέλος πάντων κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν χωρίς έχουμε κάποια αξιολόγηση για τις ε, συνέπειες ε, χρειάζεται να γίνει ανάλυση των επιπτώσεων κυρίως των κοινωνικών άρα να έχουμε και των προτέρων κάποιο είδους εις βάθος διαβουλεύσεις οπότε θα πρέπει να το αναλύσουμε και να δούμε το ότι αυτή η νομοθεσία θα πρέπει με κάθε να αποφύγει το να στρεβλώσει τη συνθήκη του ανταγωνισμού. Και θα πρέπει η εμπλεκόμενη οι οτιτοί, να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού. Οπότε κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να επιμείνω, θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Συνέπεια για όλους όσον αφορά την εφαρμογή, όσον αφορά την νομοθεσία αλλά και τη στρατηγική. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε την αναγκαία ασφάλεια δικαίου που χρειάζεται αυτό ο τομέα να δημιουργήσει τι κατάλληλε συνθήκε αυτέ που θέλει ο καταναλωτή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Τροτμάν για την έκθεσή της. Νομίζω ότι πραγματικά ανοίγει τον ορίζοντα για μια πολύ πραγματιστική και αποτελεσματική προσέγγιση στις δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Είναι μια πολύ καλή βάση για τις συζητήσει. Νομίζω όταν συζητούμε για τις τηλεπικοινωνίες συχνά σκεφτόμαστε τον τομέα αυτό καθεαυτό και λέμε ότι πρέπει να τον βελτιώσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Telecom και IT, ITC όπως είναι γνωστά. Αυτή, αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι μόνο υποδομές που μπορούν να μας δώσουν νέο δυναμικό, δεν είναι μόνο ζωτική σημασία για την λειτουργία, την αποτελεσματικότητα, την ενεργή, την δραστηριοποίηση, την ανταγωνιστικότητα όλες τις κοινωνίες είναι σημαντικότατες δοκιμασίες για τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη προκειμένου να ανταγωνιστεί άλλες περιοχές του κόσμου. Εάν δείτε τι συμβαίνει από αυτό το πρίσμα, τι συμβαίνει στο παγκόσμιο προσκήνιο, το εφιστάμενο πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες δεν έχει προσφέρει όσα θα θέλαμε. Ίσως να μην υλοποιήθηκε αρκετά γρήγορα. Ίσως να μην χρησιμοποιήθηκε ε, αρκετά όλο του το δυναμικό ίσως να μην είναι αρκετό. Όμως θα μπορούσε κανείς να πει δικαιολογημένα ότι δεν πετύχαμε όπως επιδιώκαμε. Η Ευρώπη καθυστερεί. Έχει μείνει πίσω. Όταν συζητάμε την κατάσταση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών και της αγοράς τους, μπορεί να πει κανείς, και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει, ότι έχουμε υπερβολικά πολλούς φορείς ή πολύ λίγους είναι πολλοί οι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο κάθε πελάτης χρειάζεται δύο, τρεις, άντε το πολύ τέσσερις που να ανταγωνίζονται. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι είναι πολύ δυνατοί και κάποιοι ιδιαίτερα δύναμοι. Πολύ δυνατοί στις εγχώριες αγορές τους. Άρα γίνεται πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση και οι υπόλοιποι στην αγορά αυτή. Αλλά είναι και πολύ αδύναμοι για να διατηρήσουν αμύωτο το ρυθμό της καινοτομία, την όθηση στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Είναι λοιπόν διτό το πρόβλημα. Είναι οι δύο όψεις ε, του ίδιου νομίσματος. Πολύ δυνατή, πολύ αδύναμη, πολύ λίγη, πολύ άριθμη. Και έτσι πρέπει να σκεφτούμε το τι θα πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι μεγάλο μέρος της νομοθεσίας μας κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά προστατεύει τις ε, εσωτερικές, τις εθνικές μάλλον αγορές αυτές καθ' Προκαλεί φραγμούς. Διατηρεί τα σύνορα. Όχι μόνο οι αγορές είναι εθνικές αλλά και τα συστήματα, ο συνδυασμός ε, φορέων παρεχόντων, ε, ανταγωνιστών, ε, σε εθνικών ρυθμιστών, σε κάποιο επίπεδο διατηρούν τον κατακαιρματισμό της αγοράς αυτής αυτής. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πολλοί άριθμα παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες για την πρόσβαση στην αγορά αυτή. Είναι πολλές οι στην υλοποίηση της νομοθεσίας. Ένα παράδειγμα για παράδειγμα το γεγονός ε, της ε, κατανομής του φάσματος. Είναι άνηση. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι από τη μια είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να έχουμε πανευρωπαϊκές εξελίξεις, πανευρωπαϊκή ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς, αλλά ταυτόχρονα έχουμε υπερβολικά πολλές εθνικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το ευρύ φάσμα και το τι βήματα πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε προς τη σωστή αλλαγή. Και μην ξεχνάμε ότι τα διαφορετικά βήματα πρέπει να κάνουμε πρέπει να εντάσσονται σε μια γενικότερη εικόνα. Από αυτή την άποψη, και εδώ θα ολοκληρώσω γιατί καταλαβαίνω από τις χειρονομίες της Προέδρου ότι είμαστε ήδη στο τέλος του χρόνου, θα πρέπει να διερευνήσουμε το πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερες υπερεθνικές, διακρατικές αγορές. Να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή business to business ε, συναλλαγές, αλλά μετά και business to customer. Συντονισμό στο φάσμα, άνοιγμα της ευρυζωνικότητας και πρόεδρε την διανομή σε διασυνοριακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Άντερς Δότερ, τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι με το κείμενο της κυρίας Τροτμάν. Έχει πολλές καλές προτάσεις το κείμενο. Πιστεύουμε και εμεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η κατακαιρματισμένη προσέγγιση. Η συνέπεια και η συνακτικότητα στην προσέγγιση των δικτύων βοηθούν και την νομοθεσία, του νομοθέτε μάλλον, αλλά κυρίω το κοινό και τι επιχειρήσει. Πρέπει να αποφασίσουμε σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή αγορά συνολικά. Όμω, να εκφράσω και στήριξη για κάποια στοιχεία που, ο συνάδελφο από το ΕΛΚΑ ανέφερε ε, μόνο και μόνο επειδή επιδιώκουμε τη συνέπεια και τη συνεκτικότητα του πλαισίου, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ότι θα ε, πρέπει να επιδιώκει το πλαίσιο. Και η λειτουργική, ο λειτουργικό διαχωρισμό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι ευκαιρίε που ε, προσφέρει το πλαίσιο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με του συναδέλφου για να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ εξαιρετικά ω προ τη συντομία για τα συμπεράσματα η κυρία Τροτμάν. Πρόεδρε, το συμπέρασμά μου θα είναι τάχιστο. Νομίζω ότι εδώ έχουμε έρθει για να ακούσουμε την Επίτροπο που ελπίζουμε να μας αναγγείλει και κάποιες σχετικές προτάσεις. Είπαμε ότι επιθυμούμε μια προσέγγιση συνολική, συνεπή, αλλά προσαρμοσμένη και στις ανάγκες της αγοράς, μάλιστα της ενιαίας αγοράς. Θέλουμε ανταγωνισμό αποτελεσματικό και θέλουμε καινοτομία και υπηρεσίες προς όφελος των καταναλωτών. Συμφωνώ με όλα πρέπει να αναζητήσουμε ποιοι είναι οι δυνατότεροι, ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι και πώ θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλό μίξ, ένα καλό μείγμα μεταξύ των όσων είπε ο κ. Χόκμαρτ. Το Big Bang και τα μικρά βήματα που χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι αυτή ακριβώ την ισορροπία επιζητούμε. Ευχαριστώ του συναδέλφου. Ευχαριστούμε την κυρία Τρουτμάν. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι μέχρι την 5η 11 Ιουλίου το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο που ήρθε εδώ. Ζητούμε συγνώμη για την ε, καθυστέρηση που σημειώσαμε. Επτά λεπτά. Σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας πριν την καλοκαιρινή διακοπή. Γι' αυτό και ήταν εντατική η συζήτησή μας, έντονη η ημέρα, πολύ προσκεκλημένη, πολλές εκθέσεις, πολλές ψηφοφορίες, να συγχωρείτε. Να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για την εισηγησή σας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρέπει να σας πω ότι περίμενα με χαρά αυτή την σημερινή ε, συνάντηση και χάρηκα που με καλέσατε για να μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Και βεβαίως για να ξεκινήσει έτσι πρέπει και εγώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς διακυβεύεται. Αυτό λοιπόν που επιθυμώ είναι να σας παρουσιάσω κάποιες ε, λεπτομερείς απόψεις ε, για το πώς μπορούμε να έχουμε μια διασυνδεδεμένη Ήπειρο. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ε, η ψηφιοποίηση προχωράει. Αυτό δεν είναι θέμα αν συμφωνείτε όχι. Αυτό είναι γεγονός πλέον. Έχουμε λοιπόν μια αυξανόμενη κοινή αγορά και αυτό προσφέρει προοπτικές. Εμείς αναζητάμε προοπτικές για να στηρίξουμε την οικονομία και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα πολύ βασικό ερώτημα. Τι είδους ε, μελλοντική οικονομία έχει η Ευρώπη κατά νου. Ο τομέας τηλεπικοινωνιών ε, και τα συστήματα πληροφορικής ε, δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο και αυτό με λυπεί, αλλά με κάνει και να θέλω να αγωνιστώ. Οι, οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν ε, διάφορες ε, διάφορα πρόστιμα, χρεώσεις που είναι άδικες ή χρεώσεις. Αυτά αφορούν ακόμα και τη δική μας, την κοινή αγορά. Και εγώ εξηγώ σε όλους ε, όσοι είναι έξω από εμάς ότι η κοινή αγορά είναι ένα διαμάντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει μέχρι τώρα ένας ε, χώρος που ξέρετε από την κοινή αγορά και αυτός ο χώρος είναι οι τηλεπικοινωνίες που είναι τόσο σημαντικές και συνδέονται με πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αν λοιπόν πραγματικά επιθυμούμε να υλοποιήσουμε ε, την κοινή αγορά ε, και σε αυτόν τον τομέα πρέπει να εργαστούμε. Παρεπιπτόντως, στον υπόλοιπο κόσμο σημειώνονται μεγάλα βήματα και αυτό μας επηρεάζει. Παρεπιπτόντως ε, θέλω να σας πω ότι αυτά όλα αποτελούν κίνητρα και για μας να προχωρήσουμε. Αναφέρομαι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Νότια Αμερική, η οποία μαζί με την Ιαπωνία και την Κορέα έχουν το 80% των εγγραφών εμείς έχουμε μόνο το 6% ε, και μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό έχουν ε, γρήγορο ίντερνετ. Αυτά είναι προβλήματα που αναζητούν λύσεις. Εγώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε θέλω να βρω ένα πακέτο για να τα επιτύχω όλα αυτά ε, μέχρι το Σεπτέμβρη. Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθούν τα σύνορα, ε, θα είναι πιο εύκολο να επικοινωνεί κανείς ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμενος στο υπάρχον πλαίσιο. Είναι λοιπόν σημαντικό να προχωρήσουμε σε τρεις βασικούς τομείς στη διασύνδεση. Πρώτον, για να υπάρχουν αμυγός ευρωπαϊκά δίκτυα, πρέπει να είναι εύκολο να επικοινωνεί κανείς και πέρα από τα σύνορα, χωρίς ε, να υπάρχουν ε, ασυμβίβαστοι κανόνες. Και εάν λοιπόν μπορεί κανείς να επικοινωνεί όπου επιθυμεί στην Ευρώπη, μέσα σε ένα εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τότε ε, θα πρέπει κανείς να μπορεί να επικοινωνεί όπου θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν εννοώ ε, το απλά στα λόγια, αλλά πρέπει να γίνει και στην πράξη. Να υπάρχουν εννέα συστήματα αδειοδότησης ε, με εποπτεία των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει περισσότερες ευκαιρίες να διασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο κόστος, λιγότερα εμπόδια, ακριβώς αυτό ε, σημαίνει κοινή αγορά. Και αυτό δεν είναι απλά λόγια. Αν είμαστε σοβαροί, αυτά όλα μπορούν να εφαρμοστούν και υπάρχουν ε, σε τομείς όπως ε, στις τράπεζες, στις ε, αναμεταδόσεις εκπομπών. Το μόνο που υπολείπεται είναι οι τηλεπικοινωνίες. Δεύτερον, οι πάροχοι ε, χρειάζονται ε, κίνητρα. Όσοι έχουν τα πράγματα, όλα αυτά είναι δύσκολα, κυρίως πέρα από τα σύνορα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πιο ε, συνεπείς ε, τρόποι ε, να υπάρξει τυποποίηση, πρόσβαση στα δίκτυα, αυτό που αποκαλείται Virtual Bitstream Projects και με τα σχέδια, με τα προγράμματα αυτά να διασφαλίζουμε την ποιότητα Επίσης για τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες χρειαζόμαστε κανόνες. Το διαδίκτυο η ευρυζωνικότητα ε, πρέπει να γνωρίζουν πόσο διαρκεί μια άδεια και πάρα πολλά άλλα παρεμφερή ερωτήματα. Όλα αυτά ε, θα καταστήσουν ευκολότερο να λειτουργεί ένα δίκτυο σε περισσότερες χώρες και θα μπορεί κανείς να απολαμβάνει υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας. Οι πολίτες μας πρέπει να μπορούν να έχουν ίσα δικαιώματα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ε, της ουδετερότητας. Το μπλοκάρισμα δεν είναι μόνο άδικο και ενοχλητικό για τους χρήστες, ε, κατ' ουσίαν είναι η καταδίκη και για τους ε, καινοτόμους ερευνητές. Με μεγαλύτερη διαφάνεια θα ξέρει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα του και θα είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξει κανείς πάροχο. Ε, τα επιβραβεύονται όσοι προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Αυτό είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το υπολογιστικό νέφος. Ανταγωνιστικότητα λοιπόν που θα έχει θετικά αποτελέσματα σε όλους τους πολίτες και σε όλα τα νοικοριά. Η διάδεση του διαδικτύου ε, βασίζεται στην, ε, στο στα είμαστε στην καινοτομία και θα έλεγα και σε απόλυτη ασφάλεια. Ε, για να υπάρχει καλή συμφωνία πρέπει να υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Στην <coughs> Ευρώπη δεν θα πρέπει να στοιχίζει τόσο πολύ ένα διεθνές τηλεφώνημα, όχι σε μια κοινή αγορά. Αυτά ε, θα πρέπει να γίνονται στην κοινή αγορά, χωρίς περιαγωγή. Εξάλλου, δεν πρέπει ε, να αυξάνονται οι τιμές ε, ξαφνικά και απροσδόκητα. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε <coughs> αύξηση τιμής ε, θα πρέπει να είναι αντικειμενική. Και βεβαίως σε μια πραγματική κοινή αγορά δεν υπάρχουν τεχνητές, ε, τεχνητά τέλη περιαγωγής. Αυτό εκνευρίζει. Είναι άδικο. Ανοίξει το παρελθόν. Όταν η περιαγωγή ε, είχε σχέση με σύνορα. Τώρα είναι τεχνητά όλα αυτά, δεν είναι απαράδεκτα. Και τέλος, ε, αυτό που μας υπενθυμίζει τα εσωτερικά σύνορα είναι ε, το τηλέφωνο μας που έχουμε στην τσέπη μας. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά τα παράσιτα μας το υπενθυμίζουν. Εκατομμύρια Ευρωπαίων θέλουν να έχουν καλά πακέτα στα κινητά τους θέλουν να πληρώνουν μία φορά και εκεί να συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Όχι μόνο όταν είναι στην πατρίδα τους, αλλά και όταν ταξιδεύουν. Θα πρέπει τα, το χρόνο τους ε, και τα μηνύματά τους ε, να τα παίρνουν μαζί τους όπου και αν πηγαίνουν στην Ευρώπη. Ξέρω ότι δείξατε το θέμα της ε, περιαγωγής ε, στο σχέδιο της έκθεσης, ο κύριος ε, Ρόντε, και σας συγχαίρω γιατί κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω κάτι. Δεν θα επιτύχουμε την κοινή αγορά με την απαγόρευση των τελών περιαγωγής. Το αντίθετο, με την δημιουργία κοινή αγορά θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα τέλη της περιεγωγής. Ε, οι εταιρείε έχουν όλες την ίδια πίεση να μειώσουν τα τέλη περιεγωγής, να λειτουργούν όπως είναι στην πατρίδα τους. Η αγορά θέλει να τραβήξει και να κρατήσει πελάτες προσφέροντας και δωρεάν ε, περιαγωγή. Μια αγορά λοιπόν όπου οι ε, καταναλωτές θα απολαμβάνουν τον ανταγωνισμό και όχι τα σύνορα. Εγώ έτσι θέλω να αντιμετωπίσω τη σημερινή κατακαιρματισμένη πραγματικότητα, να υπάρχει ένας, ε, μια πραγματική ανταγωνιστική κοινή αγορά. Η κατάκμηση ε, έχει ουσιαστικές συνέπειες και θα σας αναφέρω ένα και μόνο παράδειγμα. Το φάσμα. Οι χώρες δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους σχετικά με το φάσμα, αλλά ακόμα και όταν χορηγείται είναι πολύ δύσκολο, ε, είναι λοιπόν ε, αφάνταστα δύσκολο να προσφέρει κανείς ε, υπηρεσίες πέρα από τα σύνορα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να λειτουργήσουν οι κατασκευαστές, οι μηταποιητές και Γι' αυτό το λόγο το κόστος μετακυλείται στον καταναλωτή που αυτό σημαίνει υψηλότερες ε, τιμές και χειρότερες υπηρεσίες. Οι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι μεταποιητές οι οποίοι θέλουν να ανταγωνιστούν σήμερα και πρέπει να σας πω πρόσφατα κυρία Πρόεδρε ήταν ε, κυρίαρχοι σε αυτήν την αγορά οι Ευρωπαίοι μεταποιητές αυτά ας πούμε τη δεκαετία του 90 ε, και όχι μόνο σε ένα μόνο τομέα ε, όχι μόνο στα τηλέφωνα και στις ταμπλέτες πολύ σύντομα ε, θα μπορεί κανείς να συνδέσει όλες τις συσκευές μεταξύ τους που διαθέτει. Εδώ λοιπόν ε, προσφέρεται μια τεράστια επιτυχία για τους πολίτες να απολαμβάνουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ε, που υπάρχουν τη στιγμή αλλά όχι ολοκληρωμένες. Και δεν αναφέρομαι σε ένα και μόνο τομέα, αναφέρομαι γενικότερα. Ο Ευρωπαίος, ε, ευρωπαϊκός ε, τομέας ε, τηλεπικοινωνιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας και θέλω να ενισχυθεί. Ένας ισχυρός τομέας τηλεπικοινωνιών σε μια ανταγωνιστική αγορά. αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους μας και είναι γεγονός ότι η οικονομία βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία και δίκτυα. Σε τομείς από τον τραπεζικό τομέα μέχρι τα θέματα επιμελητίας και πέρα από όλα αυτά έχουμε πολλές εταιρείες που επιθυμούν διακαώς την ε, διασύνδεση που μπορεί να αλλάξει τη δουλειά τους. Θέλουν video conferencing, θέλουν υπολογιστικό νεύφος, θέλουν τρισδιάστατες εκτυπώσεις και πρέπει να σας πω ότι οι εταιρείε έχουν κουραστεί πια το να μην τα έχουν όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε και εμείς ταχύτερα. Όλοι αυτοί έχουν φιλοδοξίες στην Ευρώπη ε, και εμείς δεν μπορούμε να τους στερούμε την επικοινωνία. Σε μια οικονομία που βασίζεται στην ενημέρωση και στην επικοινωνία ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να αποδυναμηθεί πλήρως ο τομέας των ε, τηλεπικοινωνιών, ούτε να αγωνιστεί θα μπορεί, ούτε τίποτα. Δεν μπορούμε ε, λοιπόν ε, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα αυτά τα φτωχά εθνικά δίκτυα. Και αυτό παίζει ρόλο από μια ανταγωνιστική αγορά στις τηλεπικοινωνίες θα μπορούσε να αποφέρει 110 δις ευρώ το χρόνο ή σε 50 χρόνια 800 δις. Η ευρυζωνικότητα θα μπορούσε να προσφέρει 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και αυτό σημαίνει επένδυση στην ανάπτυξη. Η δική μου προσέγγιση είναι ρεαλιστική. Σήμερα τα δικτυά μας και οι κανονισμοί μας σε μεγάλο βαθμό είναι εθνικά η ρεαλιστική προσέγγιση δεν ε, σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε αυτά τα δίκτυα και να αρχίσουμε από το μηδέν. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό που έχουμε και να το προσαρμόσουμε, να ε, διαπλατείνουμε τη στενοπό, να δώσουμε ε, στις εταιρείες, τους πολίτες μια όθηση στην κοινή αγορά, καλύτερες υπηρεσίες και γνωρίζω πολύ καλά ότι εδώ και πολύ καιρό συζητάτε εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν, μία πιο ε, περιεκτική λύση όπως αυτή που ανέφερε και η κυρία Τράουτμαν ε, και βλέπω ότι η προσέγγιση της είναι ε, πολύ ελκυστική. Αλλά εγώ σας συστήνω το εξής. Να μην χάσουμε την ευκαιρία κυρία Τράουτμαν να δείξουμε την πραγματική διαφορά στην ανάπτυξη μια ρεαλιστική προσέγγιση για πλήρη αναθεώρηση ε, θα χρειαζόταν πέντε χρόνια. Και εγώ αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω για να το καταλάβουν όλοι αυτοί οι νέοι που ψάχνουν δουλειά. Δεν μπορώ να τους ε, πείσω ότι πρέπει να περιμένουμε. Το να χάνει σήμερα κανείς χρόνο σημαίνει χάνει ευκαιρίες. Ε, για δέστε λοιπόν πως άλλαξε ο κόσμος τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι εντυπωσιακό, μαγευτικό. Μιλάμε για συσκευές που δεν είχαμε πριν από πέντε χρόνια και τώρα όλα αυτά τα σκεφτούμε δεδομένα. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολύ, ενώ ε, σε άλλα μέρη του κόσμου η κούρσα τρέχει ταχύτατα. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μία άμεση παρέμβαση ώστε να έχουμε την απαραίτητη ανάπτυξη και να ε, αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό το υπάρχον πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν βήματα προς την ενιαία αγορά όπου τεχνολογία και ε, όλα μας τα μέσα θα συγκλίνουν για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της νέας πραγματικότητας. Χρειαζόμαστε ένα επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη τις δυναμικές αλλαγές που συμβαίνουν πρέπει να βρούμε το χρόνο για να τα μελετήσουμε όλα αυτά και μετά να τα εφαρμόσουμε απευθεία. Γιατί όλα αυτά είναι απαραίτητα για το μέλλον. Αλλά πρώτα απ' όλα α δημιουργήσουμε την ενιαία αγορά για τι τηλεπικοινωνίε, α λειτουργήσει αποτελεσματικά για την Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν πια εναλλακτικέ. Ε, κυρία Πρόεδρε, στην ε, θητεία αυτού ε, του Κοινοβουλίου σας δίνω ένα εργαλείο για να αποκομίσουμε μέσα ωφέλη για τους πολίτες μας και την οικονομία μας. Λιγότερη φραγμή, περισσότερη επιλογή, δικαιότερες τιμές, καλύτερες επιχειρηματικές ε, υπηρεσίες περισσότερη διαδικτύωση, περιεγωγή, ισχυρότερη οικονομία και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτά είναι τα ωφέλη της διασυνδεμένης ε, ανταγωνιστικής υπήρου. Νομίζω όλοι προς τον ίδιο σκοπό ε, εργαζόμαστε. Και εάν πιστεύετε στην Ευρώπη, πιστέψτε και στον αγώνα μας για να επιτύχουμε αυτό το αποτόλεσμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πετύχουμε μαζί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε. Είναι 17 και 54. Έχω 12 ομιλητές εγγεγραμμένου στον κατάλογο των αγοριτών, Εάν θέλουμε να μείνει λίγος χρόνος. 13 μόλις. Εάν θέλουμε να αφήσουμε 5, 5 λεπτά στην Επίτροπο για να απαντήσει, 2 λεπτά κατά κεφαλήν. Να είστε συνοπτικότατοι. 2 λεπτά για μία ερώτηση. Ξεκινούμε με την κυρία Σας eh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε κυρία Αντιπρόεδρε. Αυτή είναι η επιτροπή σας. Δεν θα επεκταθώ. Γιατί είναι αναγκαίο το να ε, αναπτύξουμε την ιστορική αγορά σχετικά με τι ηλεκτρονικέ γιατί είναι σοβαρέ οι επιπτώσει που θα έχει κάτι τέτοιο στην ανάπτυξη, την οικονομία, την απασχόληση. Ε, γιατί πάνω σε αυτά συμφωνούμε όλοι. Όλοι πιστεύουμε ότι χρειάζεται να πατήσουμε γκάζι. Και αυτό το ξέρω. Και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό το μόνο το οποίο θα ήθελα τώρα να σας πω κύριε Επίτροπε είναι ότι χρειαζόμαστε ε, να παρουσιάσετε στο Κοινοβούλιο κάτι το οποίο να αφορά την ε, νομοθετική διαδικασία για τη σημερινή συγκυρία. Πάρα πολύ ε, άμεσα μας τα είπατε, αλλά είναι πιο περίπλοκη η νομοθετική, νομοπαρασκευαστική διαδικασία εδώ στο Κοινοβούλιο από ό,τι θα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο αρμόδια, μόνη αρμόδια την Επιτροπή μας. Έχουμε συνομωδήσει και άλλες επιτροπές, αλλά τα πράγματα περιπλέγονται. Οπότε, μήπως υπάρχει κάποιο είδους πρόταση, οπότε από πλευράς διαδικασίας να είναι κάτι το οποίο να είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο. Ναι, να πατήσουμε γκάζι, αλλά έχουμε κάποια όρια, κάποιους περιορισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Επίγουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Για να δεν έχουμε κάποιο έγγραφο το οποίο πραγματικά να διακρίνεται από βιωσιμότητα, βιωσιμότητα πλευρά νομοπαρασκευαστή διαδικασία, οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα κάνουμε τίποτα παρά το ότι το επιθυμούμε. Θα πρέπει αυτό το οποίο ε, προτείνεται να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι το οποίο να είναι δόκιμο πλευρά του Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ είμαι. για την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να ρωτήσω ένα-δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, βάσει μιας πρόσφατης έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές λαμβάνουν μόνο 74% της ταχύτητας της σύνδεσης στο διαδίκτυο για την οποία πληρώνουν. Τι μέτρα προβλέπετε σε νομοθετικό επίπεδο για να προστατεύσετε τους καταναλωτές. Και σε ό,τι αφορά την προστασία του επίπεδου ευρυζωνικότητας για το οποίο πληρώνουν. Επίσης να ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες e-governance, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θεωρούνται προτεραιότητα. βάσει του συμφώνου αύξησης και μάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης. Όμως στη Συμφωνία Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για τις κατεντρίες γραμμές επί των 10 δικτύων ICT έγινε προσπάθεια να απαλληφθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών ICT. Η διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης, θα, το Connecting Europe Facility θα έχει τελικά ένα πολύ μικρό ποσό. Θα πρικοδοτηθεί με πολύ μικρό ποσό. Και εσεί ετοιμάζετε συστάσει για το Συμβούλιο του Οκτωβρίου παράλληλα. Τι μέτρα σκοπεύετε να προτείνετε προκειμένου να φροντίζετε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη να συμπεριλαμβάνει τι υπηρεσίε ICT, που είναι ζωτική σημασία για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και η τελευταία μου ερώτηση. Ε, Αναφέρεται στις νομοθετικές προτάσεις που ετοιμάζεται για την περίοδο 2013-2014. Πρόσφατα ανακοινώσατε ότι θα προβλέψετε περιπλοκότερη νομοθετική πρόταση για την άρση των τελών περιαγωγής στην εσωτερική αγορά. Ελπίζω η πρόταση αυτή να έχει λεπτομερέστερα στοιχεία για την ανάπτυξη της εσωτερική αγορά και την περιαγωγή. Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Για το 2013-2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρόντε. Ο κύριος Ρόντε. Ο κύριος Ρόντε. Η κυρία Άντρστότερ. Συνολικά είναι μεγάλη μας χαρά που η Επιτροπός θέλει ένα φιλοδόξο πακέτο για να τονωθεί η ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Όμως κάπως μας ανησυχεί το αν προσεγγίσετε τα πράγματα όπως το παρουσιάσατε, αλλάζοντας την συνοχή με το... και τη διασύνδεση με το τωρινό νομοθετικό πλαίσιο. Δείτε τι προτείνετε τώρα. Την ουδετερότητα του δικτύου. Μα το αναφέρατε και το 2009 και περιμέναμε. Περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό να γίνει. Θα ήμασταν αιώνια ευγνώμονες αν ε, γίνει η πρόταση, αλλά πολλά από τα στοιχεία που προτείνατε τώρα φαίνονται αρκετά ρηξικέλευτα. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει κάποια αποτίμηση ω προ την συνεκτικότητα κατά τη συνέπεια για το τι, το τι προτείνατε. Ιδίω γιατί τόσε πολλέ στρατηγικέ αυτή τη στιγμή ξεκινάνε ταυτόχρονα. Παντού, cloud computing και ούτω καθεξή. Νομίζω ένα από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένως είναι ότι οι πολίτες και οι καταναλωτέ μας θέλουν εμπιστοσύνη. Θέλουν να έχουν εμπιστοσύνη στην εσωτερική ψηφιακή αγορά. Για το σκοπό αυτό ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ο κατακαιρματισμό τη ε, νομοθεσία για το copyright, για τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι πολύ δύσκολο να είναι κανεί σπίτι του γνωρίζοντα όταν πηγαίνει σε μια ιστοσελίδα ότι μπορεί να παρέχεται από άλλο παρέχοντα και να ξέρει σε τι νομοθετικό πλαίσιο εμπίπτει και τι δικαιώματα θα είχε σε σχέση με αυτά που έχει στο κράτο μέλο του. Τι θα κάνει για αυτά η Επιτροπό. Όταν ε, πάω σε ένα Ιταλικό και Ισπανικό ιστότοπο, πού να ξέρω αν μπορώ να πάρω ένα παράθεμα, πού να ξέρω αν πρόκειται για ε, παράβαση κάποιας νομοθεσίας σε άλλο κάτω μέλος. Και κάτι άλλο που πολύ πρόσφατα παρατηρήσαμε. Είχαμε τα τεράστια αυτά σκάνδαλα για την κατασκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φαίνεται τα κράτη-μέλη να μην συμπαθούν το ένα το άλλο τελικά. Αυτό ε, είναι πρόβλημα και για μένα γιατί λαμβάνω πολλά ερωτήματα από τους νέους. Τι νόημα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να υποβληθούμε σε αυτό το πλαίσιο κανόνων. Ωραία θα ήταν να είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαστε. Πότε θα γίνει αυτό. Ακούω λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς οι δημόσιοι φορείς ε, της Ένωσης και των κατών μελών παρακολουθούνται από ξένου φορεί. Θα μπορούσατε αυτό τον κατάλογο να το δημοσιεύσετε. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια για τι διαδικασίε προστασία και ασφαλεία και ιδίω και τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με συγχωρείτε που με γρηγορήσα. Ευχαριστούμε ο κύριο Πρόντι. Ε, ναι. Ο κύριος Ρόντε, ε, με συγχωρείτε. Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και σας ευχαριστώ για τις φιλοδοξίες σας. Πραγματικά τις χρειαζόμαστε. Όμως, σας ευχαριστώ και για τη, τα ευγενικά σας λόγια. Ναι, όχι εγώ, αλλά εμείς, ολόκληρη η Επιτροπή, κάναμε πολύ καλή δουλειά για το ψήφισμα αυτό. Επίσης, ευχαριστώ και το προσωπικό μας το ψήφισμα έχει συνυπογραφεί από όλες τις πολιτικές ομάδες και πέρασε με μία και μόνη ψηφοφορία, με 51 ψήφους υπέρ, και καμία ψήφο κατά. Αυτό σημαίνει ότι εσείς πλέον έχετε την ισχυρότερη δυνατή εντολή που έχει δώσει ποτέ το Κοινοβούλιο για τις δικές σας τις φιλοδοξίες. Άρα είμαι πολύ ικανοποιημένο να μπορώ να πω ότι το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο και ότι έχουμε και κοινέ απόψεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο ενωμένοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Και μια άλλη ερώτηση. Τι στρατηγική χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Διότι όπως προείπα, μοιάζει τα κράτη-μέλη να μην συμπαθούν το ένα το άλλο. Το είπε και συνάδελφος, συνάδελφους, οι κυριάντες τότε. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να ξέρουμε μια στρατηγική. Και εν ώψη της Συνόδου του Οκτωβρίου. Θα μπορούσατε να πείτε ένα δυο λόγια γι' αυτό. Το σκεφτήκατε τι στρατηγική θα πρέπει να καταρτήσουμε από κοινού προκειμένου να επιδιώξουμε κάποιους από στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Ματίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ε, προκλήσεις που αναφέρατε και επίσης εκτιμούμε τις ε, φιλοδοξίες σας. Στην περίοδο την οποία διανύουμε είναι αναπόφευκτο να διερωτηθεί κανείς για τα θέματα της ασφάλειας, της προστασίας. Επίτροπε, ξέρετε τι έγινε πρόσφατα, νομίζω ότι είναι θεμελιώδου σημασία όλα αυτά. Όταν ε, βλέπουμε τι νέε προτάσει, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε και οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη στοιχεία του στο cloud, που πρέπει να ξέρουν για ποιους είναι διαθέσιμα. Είναι καθοριστική σημασία σε αυτό. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή έδωσε μια πολύ ήπια απόκριση στο σκάνδαλο PRISM. Έχει μέσα στη διάθεσή της ισχυρότατα, μπορεί να διαπραγματευτεί με τις εμπορικές συμφωνίες, ούτε αυτό το αξιοποιήσαμε, άρα υπάρχει ε, κατεπίγουσα ανάγκη διευκρίνησης. Πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ευρωπαίες πολίτησες να πιστέψουν στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα. Ε, μόνο οικονομικά ζητήματα ακούνε να, προωθούνται. Τα δεδομένα τους κυκλοφορούν ελεύθερα στο cloud. Πώς θα το εμπιστευτούν αν δεν έχουν ε, τέτοιες ε, εγγύσεις. Ήταν πολύ σαφές αυτό που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εξαιρετικό το εγχείρημα, αλλά κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να το προωθήσει. Τι θα γίνει με τα δεδομένα που δεν προστατεύονται. Μπορεί να διατεθούν στον οποιονδήποτε. Είναι καθοριστική σημασία αυτή τη στιγμή και θα σα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μου δώσετε μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κ. Ζούμπιχ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η δική μου ερώτηση αφορά ε, το εξής. Μετά το, την περιαγωγή 3 ε, πάμε στην περιαγωγή παριθμών 4 και το roaming 3 ε, θα παραμείνει ε, νομοθετικό ή η roaming 4, η περιεγωγή 4 θα επηρεάσει την περιεγωγή 3. Αυτό νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η προστασία του καταναλωτή και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω κατά πόσο όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη, όπως παραδείγματος χάνει το όριο των 50 ε, ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ερωτήματα ε, τα οποία ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ε, αφορούν το διαδίκτυο. Να μπορούν οι ίδιοι οι να επιλέξουν σε ποια χώρα ε, θα επιλέγουν πια ε, τηλεπικοινωνία. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα ε, και μπορείτε να φανταστείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει και ένα έδωσο χρηματιστηρίου όπου όλοι θα πρέπει να βάζουν τις προσφορές τους έτσι ώστε να υπάρχει και μια διαφάνεια στους ανάμεσα στους περίπου 100 παρόχους. Αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε κύριο Φανίσταροι. Ευχαριστώ. Διάβασα στην, στον τύπο πρόσφατα τις δηλώσεις του κυρίου Μπαρόζο. Η Επιτροπή Μπαρόζο 2 ε, φαίνεται να παρακμάζει. Αυτό ήταν το σχόλιο. Εγώ δεν θα έλεγα καθόλου ότι είσαστε σε παρακμή. Το αντίθετο θα έλεγα ότι είσαστε πάρα πολύ καλή φόρμα όλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα έχετε την τάση να βάζετε την τελευταία πινελιά στο μέχρι τώρα έργο σα και σε στοιχεία που είναι άκρο σημαντικά. Ήθελα να επανέλθω στο θέμα της νομοθεσίας. Τι θα πρέπει να γίνει επακριβώς, τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Γιατί έγινε συζήτηση για μια μελέτη εντυκτύπου και είμαι και εγώ υπέρμαχος της λύσης κατάργησης των τελών περιεγωγής. Γιατί να πληρώνει κανείς τέτοιες συνδρομές όταν ε, καταλήγει να καταβάλει εξωφρενικά ποσά μόλις ταξιδέψει στην Ευρώπη. Η περιεγωγή έχει μια τάση αύξησης ε, πραγματικά ε, εντυπωσιακή. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την εσωτερική αγορά και να λάβουμε υπόψη την διάσταση της απασχόλησης, την οικονομία. Θα πρέπει να ξέρουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου. Στο πακέτο που θα προκύψει θα συμπεριλαμβάνει την πρόταση για μια μελέτη αντικτύπου. Και έχετε το δίκιο τα μιλάτε για το ρυθμό με τον οποίο θα πρέπει να προχωρούμε στην υλοποίηση με τον κόσμο. Λόγω χάρη στην Κορέα του Νότου βλέπουμε. Στην Νότια Κορέα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν και εμεί προσοχή σε αυτό γιατί η αγορά μα είναι ιδιαίτερα κρυγματισμένη. Και τα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει να σταματήσουν το καθένα να βαράει το βιολί του. Διότι αλλιώ θα χάσουμε σημαντικότερε ευκαιρίε. Δεν θα τι αξιοποιήσουμε, συμφωνώ απολύτω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να διερωτηθούν πώ μπορούν να δράσουν από κοινού και να βεβαιωθούν ότι η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται και στην πράξη. Πώ μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε τι χρονικά περιθώρια. Ευχαριστούμε κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας θέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις που για μένα είναι σημαντικές σε αυτή τη φάση των συζητήσεών μας και μετά την παρουσίασή σας. Πρώτη ερώτηση. Είμαστε σε μια αγορά παγκόσμια. Η αγορά των τεχνολογιών και ε, η πόρη τη είναι ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό όσο και η ενέργεια για την ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση για τη μετάβαση την ενεργειακή ω προ τα δίκτυα, την βιομηχανία δηλαδή την παραγωγή και την ίδια την αγορά. Αλλά και το κόστο για τον καταναλωτή. Άρα πρόκειται για μια προσέγγιση σφαιρική, η οποία λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια αγορά. Έχετε για την ώρα αναφερθεί μόνο στην αγορά, με τι διασυνοριακέ διαστάσει που γνωρίζουμε. Το καταλαβαίνω και το, κατα... και το δικαιολογώ. Όλοι το επιδιώκουμε αυτό, όμω σήμερα η αγορά βρίσκεται σε φάση μετε, μετεξε, μεταλλαγής. Και χάνουμε σημαντικά μερίδια της αγοράς, διότι αν δεν έχουμε πλέον μεγάλους φορείς ή εταιρείες, το σύστημα αδειών σας, το σύστημα δικαιωμάτων, θα απελευθερώσει αστόχος την ευρωπαϊκή αγορά για μεγάλους φορείς άλλων υπήρων που θα μπορούν να κατακλείσουν την αγορά μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω την θέση σας και την οικονομική σας θεώρηση. Έχουμε μιλήσει για την Νότιο Κορέα, όμως η Νότιο Κορέα ε, οργανώθηκε και ε, χρηματοδότησε με κρατικά κονδύλια την ε, δράση της. Θέλουμε λοιπόν την οικονομική σας εκτίμηση για αυτά και κατά δεύτερον για το φάσμα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, υποστήριξα και εγώ αποφασιστικά το θέμα αυτό, υπήρξα θειασότρια Θεασότητα μάλλον, τις δράσεις της Κομισιόν υπέρ του φάσματος. Όμως θέλω να μου πείτε πώς έχουμε προχωρήσει ως προς τον απολογισμό μας σε σχέση με το παρελθόν και τη φάση 2 του πλαισίου αυτού. Και επιτά μαζί με άλλους συναδελφούς ερωτηθήκατε για το MSS. Εδώ εξεπλάγει κάπως που δεν είδα να δίνετε σοβαρή απάντηση για το πρόγραμμα αυτό. Περιμένουμε μια πρακτική απάντηση και για την ουδετερότητα του δικτύου. Να σας ρωτήσω, Επίτροπε, Πώς κατανοείτε το θέμα αυτό. Διότι δεν έχω δει ξεκάθαρα πού τοποθετήσετε. Μεταξύ απαγόρευσης οποιασδήποτε διακριτικής μεταχείρισης σε ό,τι αφορά την ε, μετακίνηση δεδομένων με τις, διακριτικές, ε, με τις διακρίσεις για, ε, λόγω στρέβλωσης της ανταγωνιστικότητας, με την ισορροπία που επιδιώκουμε για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά είχαμε 10-12 λεπτά για την έκθεση που παρουσίασα. Δύο συνάδελφοι μόνο πήραν το λόγο Χαίρομαι να μπορώ να ακούω την Επίτροπο, αλλά θα ήθελα να προσελκύσω την προσοχή σα και στο γεγονό ότι καλό είναι να υπάρχει μια ισοτιμία και ισότητα στην εξέταση των εκθέσεων τη Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πράγμα ε, το οποίο το προσέχω συνήθω, αλλά σήμερα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Συνάδελφο Έλερ, παρακαλώ. Κυρίε Επίτροπε, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο και δεν θα μακρηγορήσω. Μία πολύ απλή ερώτηση. Υπάρχει το θέμα της ε, ασφάλειας ε, και στην έκθεση λύγεται ε, λόγος ε, για οριζόντια ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις και οι τεχνολογικές λύσεις βρίσκονται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς πιστεύετε για μία πρόταση έτσι ώστε οι κανόνες διαφάνειας ε, να είναι ένα κομμάτι της αγοράς ε, που θα αφορά την επιχείρηση και τους ε, άμεσα ενδιαφερόμενους. Υπάρχει μια σχετική πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύψει στοιχείων για επιθέσεις, για την απώλεια δεδομένων σε επιχειρήσεις. Αυτά να αποκαλύπτονται στους μετόχους γιατί είναι απώλειες οι οποίες κανονικά πρέπει να αναφέρονται σε μία έκθεση. Άρα δηλαδή ε, έχουμε τις ε, ε, αποκαλύψεις στοιχείων και η πράξη περί κοινής αγοράς μας προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες. Ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τάση μας είναι να συζητάμε τα συμπτώματα της κατάτμισης ή της συνέπειας και όχι το πώς θα απαλλαγούμε αυτή τη κατάτμιση. Γι' αυτό για πέστε μας. Θα προτείνετε να ανοίξουμε αυτή τη συχνότητα. Αυτό που ζητήσει το Γενοπολί δηλαδή. Μια την πλειοψηφία. Ακόμα περισσότερο αυτή που προαναφέρατε. θα προσπαθήσετε να το κάνετε ε, με τρόπο συντονισμένο τόσο ώστε να έχουμε ευρωπαϊκά, διευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία να ε, καλύπτουν αυτό το τμήμα του φάσματος και έτσι να προλιάρουμε το έδαφος για μια πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά των διδοπλικών όσον αφορά την ε, νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Πρόκειται να εξασφαλίσετε κάποιες αλλαγές που να οδηγήσουν σε πραγματικά διασυνοριακό ανταγωνισμό, γιατί συνήθως έχουμε πάρα πολλούς α, που συναλλάσσονται στην Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί και εκεί υπάρχει ε, κατάτμιση. Οπότε χρειαζόμαστε δύο-τρεις ανταγωνιστές για κάθε περίπτωση. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να μην έχουμε προστατευτισμό των εθνικών αγορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε όσον αφορά μια νομοθεσία ανταγωνισμού. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να περιχαρακώσει τις ε, διασυνοριακές αγορές με την ισχύωση νομοθεσία και από επιχείρηση προς επιχείρηση αλλά και για τους ε, συνήθεις καταναλωτές. Μερικά από αυτά ήδη τα αντιμετωπίζουμε, αλλά άλλα απαιτούν να θεώρηση της ισχύουσης νομοθεσίας. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε για την αγορά των τηλεπικοινωνιών. Πολύ ωραία. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ και τους δύο ε, συναδέλφους που παρετήθηκαν από το να λάβουν το λόγο, Τσίτσεστερ και που σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να αφήσουμε ε, στην κυρία Επίτροπο ε, λίγα λεπτά παραπάνω για να μας δώσει απαντήσεις της. Παρακαλώ κυρία Επίτροπε. Thank you, President. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και να αρχίσω με κάτι που πρόκειψε εδώ και καιρό. Το είπατε και ορισμένοι εξημών. Για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Τις ευκαιρίες θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία γιατί τώρα υστερούμε. Καλά τα είπατε κύριε Φανίστερβα. Είπατε για Α, την κάρτα. Αυτό που έχετε στην τσέπη σας και φοβάμαι πάντα πότε θα το βγάλετε έξω από την τσέπη σας. Οπότε γι' αυτό το λόγο και αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι προσφέρεται τώρα μια ευκαιρία, όχι ένα ρήγμα α, για τους Ευρωπαίους. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σας το εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κοινωνία μας όλοι να μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την νέα ή τελος πάντων σχεδόν νέα αγορά. Κάτι το οποίο δεν είναι, θα κάνει μόνο με οικονομική δραστηριότητα, αλλά αφορά και την ηλεκτρο, το ηλεκτρονικό σύστημα υγείας την ηλεκτρονική παιδεία κλπ. επενδύσεις, ευρυζωνικότητα, υψηλή ταχύτητα στην ευρυζωνικότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ξεκάθαρο, με τρόπο συνεκτικό και συνεπή. Τέτοια αγορά θέλουμε. Και ξαναγυρίζουμε στο θέμα της ενιαίας αγοράς. Γιατί να έχουμε μια αγορά για άλλες δραστηριότητε και όχι για τα θέματά μα που συζητούμε τώρα. Άρα, να μην έχουμε φραγμούς. Ούτε φραγμούς στην είσοδο, στην ε, αγορά αυτή. Να τα πρέπει να κάνουμε. Επίσης, με ρωτήσατε Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Χάρη σε εσάς και στο Κοινοβούλιο μπορώ να πω ότι υπάρχει με τα διευθυντικά ταμεία ελπίδα. Και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε θα επιτευχθεί κάποια λύση. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά το ΣΕΦ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο και αυτό κατά κάποιο τρόπο γίνεται με αυτό το, ε, το θέμα του Connecting Euro Facility. Να απορροφηθούν έτσι αυτά τα κεφάλαια και με μόχλευση να προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα. στο Συμβουλίο του Οκτωβρίου πρόκειται να εξηγήσω τη δέσμη μέτρων που έχουμε. Καλά, όχι εγώ. Ο πρόεδρος, αλλά τόσο τη δέσμη των προτάσεων πρόκειται να εξηγηθεί τότε. Θα χρειαστούν επενδύσεις. Τώρα στον πρώτο νομοθετικό πακέτο. Όσον αφορά την πραγματικότητα, Πάρα πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο. Τόσο ώστε σε αυτή τη θητεία να περάσει η δεσμή μέλλον. Βεβαίω, βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση όσον αφορά την εξή τη κοινοβουλευτική θητεία αυτή. Αλλά χρειάζομαι την έγκριση του Κοινοβουλίου, αλλά και του Συμβουλίου. Όπω και την έγκριση του συνόλου τη Επιτροπή. Άρα θα πρέπει να γίνει ζήμωση σε όλους αυτούς τους τόσο σημαντικούς παίκτες και εμπλεκομένους. Οπότε σας οικετεύω, σας οικετεύω. Να είσαστε όσο γίνεται πιο επικοδομητικοί. Φέτος πρόκειται, πρόκειται για την ενιαία αγορά, πρόκειται για την μεθοδολογία, πρόκειται για την ουδετερότητα, πρόκειται για την βρεζονικότητα Πρόκειται για το ηλεκτρονικό διαβατήριο. Πρόκειται για την περιεγωγή. Όλα αυτά έλα συνδέονται κατά τη γνώμη μου. Ουσιαστικά είναι το θέμα ενιαίας αγοράς. Αλλά είναι και θέμα ασφάλειας όπως είπαμε. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια και τις τελευταίες ε, εβδομάδες. Το συνειδητοποιήσαμε ακόμα περισσότερο. Ότι πολλές φορές οι φίλοι μας είναι διαφορετικοί από ό,τι νομίζαμε. Και τα κλάστερ. Και το νέφος των υπολογιστών. Πάλι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω θα κρατήσει κάποιε προτάσει, κύριε Χόκμαρκ. Πάντα προσέχω. Τι εξηγείται. Θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την κατάδυμηση της αγοράς. Είναι ξεκάθαρο για μας τι πρέπει να κάνουμε. θα κάνουμε πιο εύκολη καταγγελία των συμβάσεων στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Και επίσης να είναι συμβάσεις διαφανείς. Το ίδιο ισχύει για την καταγγελία τους. Τώρα ποια είναι η σχέση μεταξύ της ε, οδηγίας εναγές και τα μέτρα που αφορούν την ε, ασφάλεια Κύριε Άντες Ντότερ, η πλατφόρμα NIS πρόκειται να συμπληρώσει την πρότασή μας και την οδηγία. Εντοπισμός κατέρης πρακτικής, εταιρείες, δημόσιο, εφαρμογή της υποχρέωσης αναφοράς κατά διαχείριση κινδύνου. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η ρύθμιση του πώς θα γίνεται η κοινοποίηση. Γιατί τώρα θα πρέπει να καλύψει όλους τους πάροχους η νομοθεσία. Έχουμε φήμη ούτως ώστε να θεσπίσουμε κάποιο ελάχιστο νομοθετικό πλαίσιο για τους παρόχους. Και αυτοί θα πρέπει να καταβάλουν πάσα ευημερία, ώστε να σεβαστούν αυτή τη ρύθμιση και να υπάρχει κάθε φορά ενημέρωση της εκάστοτε ποτικής αρχής. Με αυτές τις πρακτικές μπορεί ο ένας να οφείλει στον άλλο. Με τις εταιρείες τώρα προσπαθούμε να δούμε τι είδους ευθύνη υπάρχει και είναι περιορισμένη όταν αναφερόμαστε στις πρόσφατες εμπειρίες, τα πρόσφατα γεγονότα. Υπάρχει περιθώριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει υπηρεσίες clouding και να αναλάβει ηγετικό ρόλο και επαναλαμβάνω αυτό που λένε και οι ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία. Κάθε μειονέκτημα ή πλεονέκτημα μπορεί να αντιστραφεί. Δηλαδή το μειονέκτημα να γίνει πάντα πλεονέκτημα, αφού ενισχύσουμε τη θέση μας και προσφέρουμε ιδιωτικές και κρατικές υπηρεσίες. Προσπαθώ να πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της στρατηγικής για τον έφος και έτσι θα το συνδυάσουμε με μια ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό μπορεί να τονώσει το βιομηχανικό, βιομηχανικό κλάδο. Την επόμενη. Όχι αυτή τη εβδομάδα. Την περασμένη. Όχι την περασμένη. Την περασμένη ήμουνα σε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση υπό την Προεδρία υπό την Προεδρία του Εστονού ε, Υπουργού με εκπροσώπους από διάφορες κυβερνήσεις με θέμα ακριβώς το clouding. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι κάτι θα βγει. Σε ό,τι αφορά την περιαγωγή ό,τι αφορά την περιεγωγή από τον Ιούλιο του 2013 φροντίζουμε να επανέλθουμε στην παλιά μας υπόσχεση το roaming 3 να συμπληρωθεί από το roaming 4. Ελπίζουμε ότι αυτό που προτείνουμε τώρα θα συμπεριληφθεί στο πακέτο για την ενιαία αγορά και αν παρά το πράσινο φως από εσά και όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους τότε του χρόνου 1η Ιουλίου θα έχουμε και το επόμενο επεισόδιο του Roaming 3. Είναι σαφές. Χρειάζεται η δική σας η συμβολή, αλλά θα είναι το τελευταίο πακέτο Roaming 3. Όταν πια ολοκληρωθεί και η νέα αγορά, μπορούμε να λάβουμε και την τελική απόφαση για την αποδοχή της εσωτερικής αγοράς και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ε, πρέπει να εξελιχθεί αυτό σε ευκαιρία για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Να υπάρχει ένα υγιές ε, επιχειρηματικό πρότυπο. Δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε πλέον. Το χρονοδιάγραμμα αναφέρθηκε ήδη. Ε, the Τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright. Επαναλαμβάνομαι τώρα Λυπούμε που θα πω ότι το copyright δεν είναι καθόλου δική μου αρμοδιότητα, δεν είναι θέμα του δικού μου χαρτοφυλακίου, αλλά του αγαπητού συναδέλφου. Υποσχεθήκαμε ένα στον άλλο να ασκήσουμε πίεση μεσονομάδων που εξεργάζονται τα διαφορετικά θέματα προς ε, κάποιο αποτέλεσμα. Είναι όμω ονειρικό να το πιστεύουμε αυτό και τα όνειρα δεν γίνονται πάντα πραγματικότητα. Δεν νομίζω να μπορέσει να γίνει κάτι σε αυτή τη θητεία. Αυτό που είπατε, ένα δυο από τους όπου δεν μπορεί να εξηγηθεί στον κόσμο το τι γίνεται, ούτε μπορούμε να του δείξουμε μια ωραία ταινία σαν αναμνηστική απογενέφλια με μια ωραία υπόκρουση. Ε, δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε γιατί το να κάνουν κάτι τέτοιο στη σελίδα του στο ίντερνετ, αφού πάρουν ένα τραγούδι από όπου μπορούν από το διαδίκτυο, μπορεί να είναι παράνομο. Ε, η Ιρλανδία είναι ο ψηφιακός πρωταθλητής της Ευρώπης, με γνωστούς κινηματογραφικούς παραγωγούς, ο οποίος στην συνέλευση για τη ψηφιακή οικονομία, όπου ήσασταν πολλοί, από σας παρόντες και παρόσες, πράγμα το εκτιμώ, πρέπει να πω, είπε ότι Ωραία θα ήταν να έβγαινε η τάξη του σχολείου από το θέμα της προστασίας των πραγματικών δικαιωμάτων. Θα δίνει μια τέτοια όθηση αυτό στην εκπαίδευση, τους μαθητές, τους δασκάλους, να συζητήσουμε εάν μπορούμε να βρούμε μια-δυο εξαιρέσεις πρωτού καλύψουμε το ευρύτερο πρόβλημα που και πάλι δεν είναι ακριβώς το ζητούμενο. Ούτε πρόκειται να το λύσει η Επιτροπή Μπαρόζο 2. Νομίζω ότι μόλις το είπα, στηρίζω τα περισσότερα από τα ζητήματα που ανέφερε η κυρία Τροτμάν, θα πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον τομέα και, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα αξιοποίηση των ιδιωτικών ταμείων προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία. Ελπίζω πραγματικά ότι αν έχουμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου, αν έχουμε τη στήριξη του Συμβουλίου, θα έχουμε τη στήριξη και των συναδέλφων μου. Θα τα καταφέρουμε. Και θα είναι πραγματικά ένας τρόπος να γίνει το μέλλον μας πιο ενδιαφέρον. Αλλά δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Μόλις υποβληθεί η πρόταση θα έχετε και την ευκαιρία να αποφανθείτε. Και αυτό θα είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Πάλι θα προλάβουμε. Όπως είπε και η Πιλάρ, υπάρχουν μια-δυο διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στο Κοινοβούλιο, αλλά μαζί ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα σε μια απόφαση που θα αποδείξει ότι η οικονομία μας, οι πολίτες μας, οι επιχειρήσεις μας μπορούν να ε, ωφεληθούν και θα είναι ευγνώμονος γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Επίτροπε, εξ μέρους όλων των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλες και όλους για την συνεργασία τους τελευταίους μήνες της κοινή μας δουλειάς. δουλειάς. Ευχαριστώ τη γραμματεία, τους συνεργάτες μας, ευχαριστώ τους και τις διερμηνείς. Θα ξαναβρεθούμε στις 2 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνεδρίαση πριν την καλοκαιρινή διακοπή. Ε, κοιτάξτε να περάσετε καλά γιατί μετά έχουμε ένα εξάμεινο εντατικών εργασιών. Ευχαριστώ και καλές διακοπές.